Uh, Καλησπέρα σε όλους. Ας ξεκινήσουμε. Έχουμε ακρόαση. Impact and... Για τις συνέπειες του Brexit, τον αντίκτυπο του Brexit στη διοίκηση της Ουαλίας, Σκοτίας, Βορείου Ιρλανδίας και στην υπεράκτια κτήση του Γιβρατά. Διάφορες διαστάσεις του Brexit. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χαίρομαι που καλωσορίζω δύο εμπειρογνώμονες. Τον Τζόναθαν Τόγκ, το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Θα μιλήσει πρώτο. για τον αντίκτυπο και συνέπειε του Brexit στη Βόρεια Ιρλανδία και ο Μάικλ Κίτινγκ, καθηγητή Μάικλ Κίτινγκ από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν για τι συνέπειε του Brexit στο Γιβραλτάρ ε, και τι αυτόνομε περιοχέ σκοτία τη Ουαλία και τη Βορείου Λοιπόν, έχετε το λόγο καθηγητά Είναι εκτός μικροφώνου. Thank you very much indeed. Uh, I'm very... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσω ένα τεταρτάκι, 20 λεπτά. Θα περιγράψω κάποια θέματα. Τα οποία επηρεάζουν την Βόρεια Ιρλανδία ιδιαίτερα. Εκεί που υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιρλανδικής, ε, Βρετανικής ενωτικών εθνικιστών και λοιπά, Συμφέιν όλων των φορέων της Βορείου και της Ιρλανδίας είναι ότι η Βόρεια Ιρλανδία, είναι ότι η Βόρεια Ιρλανδία πειράζεται περισσότερο από το Brexit και κυρίως αρνητικά επηρεάζεται από το Brexit. τοσα 15-20 λεπτά δεν μπορώ να προτείνω λύσεις, αλλά να σκεγγραφίσω ε, διεξόδους προς εξέταση. Το βασικό θέμα έχει αναφερθεί εκτενώς. Τα βασικά θέματα έχουν αναφερθεί, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πώς θα αντιμετωπιστούν. Το προφανέστερο, και το κρατήσουμε για το τέλος, είναι τι γίνεται με τα σύνορα στην ίσο της Ιρλανδίας, στα πλαίσια της Θελωνιακής Ενώσεως και των κοινών εξωτερικών δασμών. Αν δείτε τι γίνεται Νορβηγία, Νορβηγία Σουηδία, Γαλλία, Ελβετία, στα σύνορα αυτά, υπάρχουν τελωνιακά καθεστώτα και στα δύο σύνορα και το ερώτημα προκύπτει πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τελωνιακό καθεστώς και αναζωγόνηση σύνορων, διότι υπάρχουν πολιτικές ευαισθησίες σε αυτά τα σύνορα. Πώς μπορούν να αποφευχθούν στην Ιρλανδία. Μετά ίσως κάτι λησμονήθηκε. Ο βαθμός των συνεισφορών ε, της Βρετανίας, ε, της Βορείου Ιρλανδίας στο Βασίλειο. Πολύ μεγάλο ποσοστό εξαρτάται από την Βρετανία. Θα πληγεί περισσότερη η Βόρειο Ιρλανδική. Μάλλον εξαρτάται πολύ από τι επιδοτήσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και θα πληγεί πολύ. Δεν θα μιλήσω τώρα στην συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή και πώ θα πρέπει να διατυπωθεί σε κάποια μορφή. Τι μορφή θα πρέπει να έχει. Και άλλε στοιχείε που θα ήθελα να τονίσω ο Ποια είναι η ταυτότητα Ιρλανδική ε, των εθνικιστών στη Βόρεια Ιρλανδία που εγγυάται η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και ο διχασμός, η διέρεση που υπάρχει στη Βορεια η Δεν μπορεί η διοίκηση της κα, έχει καταρρεύσει το από τον Ιανουάριο και μόνη φωνή που ακούγεται είναι από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον υπεύθυνο ε, για τη Βόρεια Ιρλανδία. Λοιπόν, τα αποτελέσματα στη βορεια σε αυτό το Brexit βλέπετε ότι είναι κάπως διαδική αντιμετώπιση. Καθολικοί, ε, προτεστάτες κλπ. Αυτοί που θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Αν είσαι καθολικός, αν είσαι εθνικιστής, αν θεωρείς τον εαυτό σου Ιρλανδό, τα ποσοστά εκείνων που θέλουν να μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλά. Αν είσαι προτεστάντη στη Βόρεια Ιρλανδία, αν είσαι ενωτικός, ή αν θεωρείς τον εαυτό σου Βρετανό. Και αυτό δείχνει την πολιτική αστάθεια στη Βορειοελλανδία και αυτές οι διαφορές δεν είναι συμφιλιώσιμες, διότι δεν μετανιώνει καμία πλευρά για τη θέση της. Αν δείτε τη διαφάνεια εδώ, το δημοψήφισμα του Brexit. Ποιο πολιτικό κόμμα ε, το υποστήριξε στη Βόρεια Ελλανδία. Ξεχάστε το TUV που είναι μικρό κόμμα αριστερά. Δείτε τα βασικά κόμματα, το TUP, το Δημοκρατικούς Ενωτικούς, που εκπροσωπεί κυρίως τους προτεστάντες στη Βόρεια Ιρλανδία, 70% των υποστηριχτών του κόμματο αυτό υποστήριξαν αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η θέση είναι αμετάβλητη. Λοιπόν, έχουμε τα πορίσματα του 2017 και τη μελέτη που έκανε το Συμβούλιο για κοινωνικά και οικονομικά θέματα και η θέση δεν άλλαξε. Μεταξύ των υποστηριχτών του DUP ε, θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Sinn Féin που εκπροσωπούν ε, τους καθολικούς εθνικιστές στο Βορρά, 86% υποστήριξαν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το στοιχείο στις γενικές εκλογές έφτασε στο 90%. Οπότε έχει αυξηθεί ο διχασμός η διαφορά στην, ε, στη Βόρεια από το Brexit. Έχει τροφοδοτήσει την πολιτική αστάθεια. Δεν είναι ο μόνος λόγος που ε, κατέρευσαν η πολιτική θεσμοί εκεί, αλλά τροφοδότησε και αύξησε την ε, πολιτική αστάθεια που χαρακτηρίζει τη Βόρεια Δεν έχουν αλλάξει θέσεις από καμία πλευρά. Αυτά που βλέπετε είναι από το DUP και το μανιφέστο του DUP στις πρόσφατες εκλογές όπου είπαν ότι είναι σωστό να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που υπάρχουν στοιχεία ότι οικονομικός πώς ο αντίκτυπο για τη Βόρεια Ιρλανδία θα ε, είναι αρνητικό και επιζήμιος. Αριστερά στη διαφάνεια βλέπετε με κόκκινο τι περιοχέ εκείνε των ενωτικών στη Βόρεια Ιρλανδία στι γενικέ εκλογέ, στι εκλογέ που έγιναν και πράσινα του εθνικιστές στη Βόρεια Ιρλανδία, τι περιοχέ του. Βλέπετε αυτό το διαδικό, αν θέλετε, διχασμό που τονίστηκε περισσότερο ε, από τη διαίρεση, το διχασμό όσον αφορά την τοποθέτηση για τον Brexit. Τώρα, πώς θα λυθούν τα προβλήματα της Βόρειας Ιρλανδίας. Σταθώ αυτό που θα έπρεπε να είναι εύκολο και το μόνο θέμα που μπορεί να επιληθεί εύκολα, ποικιλοτρόπως. Ο κοινό χώρο ταξιδίων, διμερή διευθέτηση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Ελευθερία διακίνηση άνευ ελέγχων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδία. Τι πρέπει να πούμε, ότι προηγήθηκε της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προχρονολογήθηκε, η διευθέτηση αναγνωρίζεται σαν κάτι νόμιμο την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται στο πρωτόκολλο 20, άρθρο 2 της συνθήκης της Λισαβόνας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Καμία χώρα δεν θέλει να ε, σταματήσει αυτό το χώρο. Αν δείτε την κλίμακα των διελεύσεων των συνόρων που υπάρχουν εκεί μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας Ιρλανδίας, συνήθισε ο κόσμος επί σειρά δεκαετιών τον κοινό αυτό χώρο διακίνησης και δημιουργείται το ερώτημα αυτή η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα διατηνόμουν ότι αυτό μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα, οπότε ο κοινό χώρο του ταξιδίων μπορεί να παραμείνει. Με τη διακίνηση μπορεί να διατηρήσει έτσι την κινητικότητα των ανθρώπων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδία και Δημοκρατία Ιρλανδία, πιο συγκεκριμένα πιο δύσκολα θέματα τώρα που ξεπερνάνε τον κοινό αυτό χώρο διακίνησης ταξιδιών και σχετίζεται με την Ευτική Συμφωνία του 1998 τη Συμφωνία Μεγάλη Παρασκευή για τη Βόρεια Ιρλανδία. Και εδώ τα πράγματα περιπλέκονται, διότι η Συμφωνία Μεγάλη Παρασκευή στην καρδιά τη εμπεριέχει την ίση νομιμότητα των δύο παραδόσεων που ισχύουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Καθολικούς ενωτικούς και τους προτεστάντες Λοιπόν, η συμφωνία δίνει σαν εγγενετής δικαίωμα την Ιρλανδική ηθαγένεια σε εκείνου που γεννήθηκαν στο νησί τη Ιρλανδίας. Εκείνοι που ήθελαν μπορούσαν να είναι Ιρλανδοί υπήκοοι. Άρα θα παραμείνουν κατά κάποια μορφή πολίτες Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αυτή θα γίνει τη Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Πώς θα αναγνωρίζεται από εκείνου που θεωρούν σε αυτού του Ιρλανδού. Και είναι περίπου εξίσου αυτοί που θεωρούν ότι είναι η Ιρλανδία, όπω και αυτοί που θεωρούν ότι είναι Βρετανοί, εντό τη Βορείου Ιρλανδία μετά την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και εγώ έχω τονίσει δύο επιλογέ. Δεν είναι πολύ καλέ, δεν είναι ικανοποιητικέ για να καλύψουν το θέμα αυτό τη διατηρήσεω ε, τη Ιρλανδική υπηκότητα και τη υπηκότητα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα, να δώσουν στου Ιρλανδού πολίτε στη Βόρεια Ιρλανδία το δικαίωμα να ψηφίζουν στι ευρωεκλογέ. Μετά, τι γίνεται αυτοί θεωρούνται σαν Ιρλανδοί που μπαίνουν στον Ιρλανδικό πληθυσμό και στις έδρες που κατανέμονται και δίνονται στην Ιρλανδία, οι ενωτικοί θα έχουν αντίρρηση να υπάρχει άλλο ένα κυρίαρχο κράτος που επιτρέπει σε πολίτες που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να ψηφίζουν σε εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο όταν ζουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά κάπως έτσι αναγνωρίζει κανείς τη διπλή αυτή ηθαγένεια ε, την Ιρλανδική με τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις. Αλλιώς πώς θα αναγνωριστεί και θα προστατεύεται, διότι στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής υποτίθεται ότι θα διατηρεί και η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μετά έχουμε τη συμφωνία αυτή καθεαυτή της Μεγάλης Παρασκευής. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα με τη συμφωνία είναι η πρώτη ομάδα. Ε, πώς δίνονται εξουσίες στη Βόρεια Ελλανδία, διάφορες αρμοδιότητες και πώς τα και να μοιραστούν εξουσίες μεταξύ των ε, εθνικιστών και των ε, ενωτικών. Και εκτο αν το κρύβουν τα κόμματα, δεν υπάρχει κάποια προοπτική να επιστρέψουν σε αυτό, στο μοίρασμα των εξουσιών στη Βόρεια Ελλανδία. Αλλά τότε γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση συναρτήσει τη συμφωνία αυτής. Πάμε τώρα στην Ιρλανδική διάσταση, στο δεύτερο, στη δεύτερη πτυχή και παραθέτω κάποια πτυχία, κάποια κομμάτια κειμένου που μας αφορούν. Αναφέρεται εκπροσώπηση ε, της, ε, της Ιρλανδικής διαστάσεως συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ενωμένης Ιρλανδίας και της εφαρμογής της, ε, ε, των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίσο της Ιρλανδίας τις απόψεις του Υπουργικού Συμβουλίου Βορρά Νότου που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα λαμβάνει την υπόψη η Ευρωπαϊκή Πολιτική εντός του Υπουργικού ε, Συμβουλίου Βορρά Νότου. Πώς θα παραμείνει αυτό αν είναι εκτός του Ευρωπα... Ευρωπαϊκής Ενώσης του Ηνωμένου Βασίλειου. Το βάρος θα πέσει στου ώμου τη Ιρλανδική κυβερνήσης όσον αφορά την ε, πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και το Ηνωμένο Βασίλειο τι θα κάνει όσον αφορά την πολιτική του. Δεν είναι να κανεί από το τι... να σβήσει κανεί διάφορε φράσει είναι μια διεθνή συνθήκη που έχει καταχωρηθεί στον ΟΗΕ. Μπορεί να συμφωνηθεί διμερό μεταξύ των κυβερνήσεων Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ετέθη όμω το δημοσίφισμα συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή ε, στην ίσο τη Ιρλανδία, σε βορρά και νότο. Εάν αλλάξει η συμφωνία αυτή, θα πρέπει να τεθεί δημοψήφισμα παρομοίω, να υποφύσει σε δημοψήφισμα, ή θα προχωρήσει η κυβέρνηση και θα αναδιατυπώσει τη συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή χωρί την νομιμότητα που θα χορηγείται από τους λαούς που διαμένουν στην ίσο της Ιρλανδίας. Αν θεωρείτε αυτά είναι δύσκολα, mm. πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Η σημασία εμπορικών σχέσεων με την ίσο της Ιρλανδίας, στο σύνολό της. 60% των εξαγωγών της Βορείου Ιρλανδίας πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγαλύτεροι αποδέκτες του εμπορίου είναι η Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Βέβαια δεν είναι αρχή και το τέλος γιατί η Βόρεια Ιρλανδία έχει πολύ περισσότερο εμπόριο. Ε, εμπορεύεται με πολύ περισσότερο με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Μεγάλη Βρετανία. Πέρα από τι εξαγωγέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεγάλο πελάτη είναι η Ιρλανδική Δημοκρατία τη Βορείου Ιρλανδία. Άρα, ερώτηση. Τι θα συμβεί στα σύνορα. Όσον αφορά την άνευ το άνευ εμποδίων εμπόριο που διέρχεται τα σύνορα όταν αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιοι τομεί είναι βάλωτοι. Η γεωργία καταρχά είναι βάλωτη, διότι η κλίμακα των δασμών, αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο άνευ συμφωνία, θα επηρεάσει το εμπόριο. 57% για εξαγωγέ γάλακτο, 40% για τυρί, ε, θα πέσουν αυτοί οι δασμοί στι εξαγωγέ Βορείου Γεωργία, 35% των εξαγωγών τη Βορείου Πολύ πάνω από το επίπεδο που είναι αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μεγάλο εισόδημα από τα, για τα αγροκτήματα προέρχεται από την ΚΑΠ. 60%, μπορεί να φτάσει και 80%. Πρέπει να τονιστεί λοιπόν ότι πολλοί γεωργοί ψήφισαν να αποχωρήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση η ταυτότητα καμιά φορά επικρατεί των οικονομικών, υπερισχύει των οικονομικών στη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά ο πρώτος, ο υφυπουργό, ο αρμόδιος, ο, μάλλον ο αντιπρόσωπος κυβερνήσης της Βορείου Ιρλανδίας είπε ότι είναι πολύ ευάλωτη η Βόρεια Ιρλανδία όσον αφορά την ε, απώλεια χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την επιβολή δασμών στα αγαθά της. Υπάρχει κάποια λύση μετά από αυτή τη ζωφερή εικόνα που προέρχεται από τα στοιχεία και παρουσίασα. Ποιε είναι οι δυνατότητε που υπάρχουν. Προσπάθησα να παραθέσω κάποιε δυνατότητε. Πολιτικό πώ είναι πολύ ευαίσθητα κάποια από αυτά τα σημεία και ενδεχομένω ε, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Όμω πρέπει να εξεταστούν όλα τα σημεία σε κάποιο βαθμό. Πρώτα απ' όλα, το Ηνωμένο Βασίλειο στο σύνολό του, ενώ είπε θέλει να αποχωρήσει από την ενιαία αγορά και την Τελωνιακή Ένωση, αντιστρέφει το θέμα της Τελωνιακής Ενώσεως στη θέση του που περιγράφεται στο έγγραφο τοποθέτησης και πληρώνει για πρόσβαση στην Τελωνιακή Ένωση να μην υπάρχουν δασμοί και να, διατηρηθεί, να διατηρηθούν ήπια σύνορα των ΣΥΠΗΝ, να μην υπάρχουν δασμοί, κανόνες περί καταγωγής, προελεύσεως κλπ. Το Ηνωμένο Βασίλειο στο σύνολό του συναλλάσσεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα ικανοποιεί την Ιρλανδική Δημοκρατία και το δέχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, κανόνε προελεύσεως, δασμοί και κανόνε ε, που ταιριάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, αν αυτό είναι εφικτό, γιατί να δώσει αδοσμολόγητε ε, δυνατότητα εμπορίου άνευ δασμών η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Βασίλειο κατά παραγγελία όπω το βολεύει. Επόμενη επιλογή. Ειδικό καθεστώ για τη Βόρεια Ιρλανδία δεν χρησιμοποιούν το όνομα αυτό, διότι οι ενωτικοί δεν θέλουν ένα ειδικό καθεστώ για τη Βόρεια Ιρλανδία. Πιστεύουν ότι ειδικό καθεστώ στη Βόρεια Ιρλανδία τη βάζει στα, στη, στις του Ηνωμένου Βασιλείου και σιγά σιγά μπορεί να γλιστρήσει προς μια Ενωμένη Ιρλανδία που είναι κατάρα για τους ενωτικούς. Και στηρίζονται οι εθνοτικές θέσεις, αυτές που περιγράφονται από το Sinn ειδικό καθεστώ τελωνιακό για τη Βόρεια Ιρλανδία, άρα δοσμολόγει το εμπόριο στην ίσο της Ιρλανδίας, αυστηροί κανόνες για το τι μπορεί και δεν μπορεί να στείλει στην υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε θα υπάρχει ένα είδο δασμών για την υπηρετική Βρετανία που θα ενοχλεί τους ενωτικούς, αλλά όλη η Ιρλανδία τελικά θα διέπεται από ελεύθερο εμπόριο και η Βόρεια Ιρλανδία θα μείνει στην πράξη μέλος της Τελωνιακής Ενώσεως. Είναι μια λύση. Πολιτικά όμως είναι ε, πάρα πολύ δύσκολο να το πουλήσει στους ενωτικούς. Κυρίως ο όρος ειδικό καθεστώς είναι δύσκολος. Ποιες άλλες ε, λύσεις έχουμε. Διάφορες διμερεί τομεακέ συμφωνίε μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκή Ενώσης που θα καλύπτει τις εξαγωγές της Βορειοελλανδίας, κυρίω στη Γεωργία. Είναι μια λύση αυτή. Παραμένουν ήπια σύνορα, μαλακά σύνορα, διότι δεν επιβάλλονται μεγάλοι δασμοί όσον αφορά το εμπόριο, δεν επιβάλλονται δασμοί στα περισσότερα προϊόντα που διέρχονται τα σύνορα. Άρα δεν χρειάζεται ένα τελωνιακό καθεστώ. Άλλη επιλογή. Έχει δασμού, αλλά εξασφαλίζει ότι έχεις μαλακά σύνορα. που Όλα τα πολιτικά κόμματα λένε ότι όλοι θέλουν αυτά τα σύνορα. Και οι ενωτικοί θέλουν, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει, η ελληνική κυβέρνηση θέλει. Δεν μπαίνει κανένα μηχανισμό τελώνιακο κοντά στα σύνορα ελέγχων. Είτε γίνονται στο διαδίκτυο ή μακριά από τα σύνορα οι έλεγχοι. Διότι υπάρχουν μεγάλε πολιτικέ ευαισθησίε όσον αφορά αυτά τα συγκεκριμένα σύνορα. Άρα, τελωνιακό καθεστώ είναι σκληρό το Brexit, αλλά η δράση τελωνιακή δεν λαμβάνει χώρα εκεί που είναι ευαίσθητα τα πράγματα, στα σύνορα. Είναι κάτι βιώσιμο, υπάρχουν τεχνικές λύσεις σε ένα πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχουν σημαντικά ερωτηματικά όσον αφορά αυτό. Τελική επιλογή. Κάτι ανέφικτο, πιθανότατα, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχουν τελωνιακά καθεστώτα δασμοί, ρυθμίσεις όλα γίνονται βάσει εμπιστοσύνη. Τα δύο βασικά αγαθά που περνάνε ελαφριά από τα σύνορα είναι ο καπνό και τα καύσιμα. Σύμφωνα με τι αστυνομικέ υπηρεσίε τη Ιρλανδική Δημοκρατία και τη Βορείου Ιρλανδία, αυτά τα δύο αγαθά από μόνα του ε, έχουν ελαφρεμπόριο ύψου πολλών εκατομμυρίων. Άρα θα ήταν αφελές να υποθέσουμε ότι αυτή η τελική ε, επιλογή θα ήταν βιώσιμη αν υπάρξει hard Brexit, σκληρό Brexit, θα υπάρξει κάποια, κάποια τελωνιακή δράση. Άρα πού θα γίνονται οι έλεγχοι τελωνιακοί, σε ποιο σημείο. Κλείνοντας, λόγω χρόνου, υπάρχουν πολιτικές επαισθησίες στα σύνορα. Μεγάλες. Και είναι το πιο σημαντικό θέμα, το σημαντικότερο πρόβλημα όσον αφορά το Brexit και επηρεάζει τον ΕΒ, το λέω εγώ, η Τερέζα Μέη στο δημοψήφισμα στην εκστρατεία είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να, παραμείνει, να παραμείνουν τα σύνορα τα ίδια. Πώς θα ήταν δυνατόν να παραμείνουν ίδια τα σύνορα αν έχει τη μία πλευρά εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την άλλη πλευρά εντός. Είναι κάτι που δεν εξετάστηκε, δεν λύθηκε μετά από ένα χρόνο. Δεν λέω ότι η επιστροφή στα κανονικά σκληρά σύνορα θα οδηγήσει σε μια επάνωδο της βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά πρέπει κανείς να το εξετάσει. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της βίας εντελώς στη Βόρεια Βλέπετε τα στοιχεία της αστυνομίας της Βορείου τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπάρχει σοβαρό επίπεδο απειλή. Δεν θέλω να είμαι ο πρώτος που προσπαθεί να ενσταλλάξει ε, την ιδέα ελέγχου τελωνιακού στα σύνορα. Εάν εκεί καταλήξουμε. Υπάρχει πρόβλημα. Οξύ. Πρέπει να λυθεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Professor Tang. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κίτιν, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Η δικιά μου εργασία ασχολείται με το θέμα της Σκοτίας, της Ουαλίας και του Γιβραλτάρα. Συμπληρώνει κάποια από αυτά τα οποία είπε ο Τζον, αλλά υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία που δεν ανακύπτουν στις άλλες επαρχίες και αντιστρόφως. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στην σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος και της αποκέντρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά κάποια συγκεκριμένα πράγματα για το τι προκύπτει από το Brexit και την μέχρι τώρα διαδικασία και την ε, κοινοποίηση του άρθρου 50. Πρώτα απ' όλα έχουμε την φύση την κρατική του Ηνωμένου Βασιλείου και την σχέση με την υπερθνική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές φορές λέμε ότι το Brexit αφορά την επαναφορά της κυριαρχίας ε, στον Βρετανικό λαό και στο Βρετανικό ε, Κοινοβούλιο ως εάν να ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο ένα ενιαίο εθνοκράτος. Βλέποντας όμως την κατάσταση εκτός Αγγλίας από τα άλλα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια περίπλοκη πολυεθνική ένωση, στην οποία το κάθε έθνος έχει διαφορετική σχέση με το κέντρο και πιθανώς και με την Ευρώπη, την οποία η κυριαρχία είναι κοινή και οι άνθρωποι έχουν πολλαπλέ ταυτότητε. Ξέρουμε ότι στη Σκοτία περισσότεροι αισθάνονται Σκοτσέζοι και Βρετανοί και βεβαίω ε, το ποσοστό θα έλεγα μεταξύ των δύο διαφέρει. Γιατί όλοι έχουν αυτέ τι πολλαπλέ ε, ταυτότητε και παρόμοια πράγματα ισχύουν και στην Ουαλία. Βεβαίω, ε, αν το δούμε έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο και ως ένα σύνταγμα το οποίο εξελίσσεται ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια με μια σταδιακή διαδικασία αποκέντρωσης προς τα μικρότερα έθνη. Μια διαδικασία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της Αγγλίας της ίδιας, αλλά έχει προχωρήσει στην Σκοτία και την Ουαλία και προχωρήσουμε και αν δούμε ότι προχωράμε προς ένα ιονί ομοσπονδιακό σύστημα που δεν έχει αυτό το όνομα και πηγαίνουμε προς μια άγνωστη κατεύθυνση. Εάν λοιπόν δούμε έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε μοιάζει πολύ με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό η ευρωπαϊκή αυτή διαδικασία της αποκέντρωσης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και οι δύο διαδικασίες έχουν πάει χέρι-χέρι. Γι' αυτό ακριβώς η αφαίρεση του ευρωπαϊκού πλαισίου δημιουργεί προβλήματα. Ένα άλλο γενικό σχόλιο είναι ότι η ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε να έχουμε μια πολύ πιο εκτεταμένη αποκέντρωση από ό,τι θα ήταν δυνατή αλλιώς. Γιατί υπάρχουν βεβαίως ακριβώς τα ευρωπαϊκά προβλήματα, τα οποία τα ευρωπαϊκά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζει ζητήματα ανταγωνισμού, περιβάλλοντος κτλ. Οπότε σε πολλά πράγματα δεν υπάρχει βρετανική πολιτική, δεν υπάρχει βρετανικό πλαίσιο και δεν υπάρχει βρετανικό υπουργείο. Αυτό περιλαμβάνει την εκπαίδευση, το οποίο εντάξει δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για την Ένωση, αλλά περιλαμβάνει και τη γεωργία, το περιβάλλον, σημαντικά τμήματα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών και στους τομείς αυτούς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κοινούς μηχανισμούς μόνο εντός της Ευρώπης. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί για να καθορίζουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στην κοινή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ασύνηθες μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης ε, γιατί δεν είναι ομοσπονδιακό κράτος το Ηνωμένο αλλά δεν είναι και κεντρικό κράτους. Οπότε, εάν δεν υπάρχει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχουμε διάφορες δυσκολίες που ανακύπτουν από το Βρετανικό Σύνταγμα και έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία προτιμούσαμε μέχρι τώρα να μην θίξουμε γιατί δεν θα συμφωνούσαμε στο αποτέλεσμα. Κάπως σαν το θέμα της Βορείας Ιρλανδίας όπου έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία βεβαίως δεν τα εξτομίζουμε και οπωσδήποτε μέχρι στιγμής η Ευρώπη μας διευκολύνει. Τέλος υπάρχει μια ρήτρα σε όλες τις ρυθμίσεις περί αποκέντρωσης που λέει ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο ισχύει απευθείας. Τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και το ίδιο ισχύει για την ΕΣΔΑ, τη Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έτσι ώστε το κοινό πλαίσιο προέρχεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα γίνει αυτόματα μετά το Brexit. Κάτι πρέπει να γίνει και το ελάχιστο που θα γίνει είναι να φύγουν αυτές οι ρήτρε που λένε ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις πρέπει να ακολουθούν το ευρωπαϊκό δίκαιο γιατί δεν θα υπάρχει πια ευρωπαϊκό δίκαιο στο Ηνωμένο Βασίλειο οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Και εκεί βρίσκεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν διαφορετικό. Η Βόρεια Ιρλανδία μας είπε ότι ε, η πλειοψηφία ήταν υπέρ της παραμονής, αλλά με διαφορά μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Στην Σκοτία το αποτέλεσμα ήταν 62% υπέρ της παραμονής, που είναι ουσιαστική διαφορά και στην Ουαλία το αποτέλεσμα ήταν επίσης παρόμοιο με της Αγγλίας και πάντα υπάρχει βεβαίως και διαφοροποίηση εντός της Αγγλίας αλλά οι δύο αυτές ψηφοφορίες σε Βόρεια και Σκοτία υπέρ της παραμονής μπορεί να μην είχαν κάποιο άμεσο αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα αλλά έχουν εξαιρετική πολιτική σημασία και επηρεάζουν και την διαπραγματεύση. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα συμβεί. Υπάρχει σύγχυση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχουμε γραπτό σύνταγμα. Έχουμε κάποιους νόμους ε, που αφορούν την αποκέντρωση, αλλά είναι κοινή νόμη, αλλά βεβαίως υπάρχουν κάποιες συμβάσεις ε, και ουσιαστικά λένε ότι οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων νομοθετικών σωμάτων δεν θα αλλάξουν χωρίς ε, την συνένεσή τους. Ε, δεν είναι δεσμευτικό, είναι όμως μια σύμβαση που υπάρχει και θα λέγαμε ότι έχει βάση στο Βρετανικό Σύνταγμα. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι το ένας απλός τρόπος για να λυθούν τέτοιες διαφωνίες και οπωσδήποτε τα δικαστήρια δεν είναι σε θέση να κάνουν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό καταλήγουμε, θα καταλήξουμε σε κάποιες συνταγματικές σύγκρουσεις. Τα σενάρια λοιπόν που ίσως προκύψουν ε, είναι κατανοητά στο πλαίσιο τριών κεφαλαίων κάθε ένα από τα οποία βεβαίως περιέχει συγκεκριμένα προβλήματα. Το Brexit θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν εκ νέου συγκεντρωτισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν π.χ. επανέλθουν αρμοδιότητες στο Westminster από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω αυτό είναι γνωστό στην Σκοτία και την Ουαλία, αλλά ε, όχι τόσο στο Λονδίνο γιατί ε, αντιλαμβάνονται διαφορετικά το κράτος και πολλοί στα Υπουργεία του Λονδίνου θεωρούν ότι επαναπατρίζουμε τις αρμοδιότητες, ενώ στη Σκοτία και την Ουαλία λένε «Ε, πού θα πάνε αυτές οι αρμοδιότητες και εξουσίες. Το θέμα και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν περισσότερο είναι αυτά τα οποία είναι υποκεντρωμένα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Π.χ. η γεωργική πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική, 99% ε, σε αυτές τις περιπτώσεις και όπως είπα κάποιες πτυχές δικαιοσύνης και εσωτερικών. Υπάρχει μια ευρεία συμφωνία στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους πλαίσιο για αυτά τα πράγματα, κάποιος συντονισμός που θα αντικαταστήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχουμε φτάσει στο σημείο που η Βρετανική, η Σκοτσέζικη και η Ουαλική κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει. δεν έχουν συμφωνήσει το πώς θα γίνει βεβαίω. Το Ηνωμένο Βασίλειο στο σχετικό νομοσχέδιο προτείνει όλες αυτές οι αρμοδιότητες να επανέλθουν στο βρετανικό επίπεδο και κατόπιν το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποφασίσει ποιες αρμοδιότητες μπορεί να εκχωρήσει η κυβέρνηση Σκοτίας και Βαλίας λένε πραγματικά πως αυτό είναι απαράδεκτο, ότι είναι δικέ τους αυτές οι αρμοδιότητες και όχι του Westminster. Είναι ένα θέμα αρχής και έχουν πει ότι δεν θα προτείνουν ε, στις εθνοσυνελεύσεις τις αντίστοιχες να συνενέσουν σε αυτόν τον νόμο. Τι θα γίνει λοιπόν αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν το ξέρουμε. Πιθανώς νομικά τίποτα, αλλά και πάλι Βεβαίω, έχουμε τις συμβάσεις αυτές οι οποίες δοκιμάζονται και μπορεί να οδηγηθούμε σε μια αντιπαράθεση για το πώς ακριβώς θα εγκριθεί αυτός ο νόμος και αν χρειάζεται την έγκριση όλων των εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου και μετά κάπως ευρύτερα η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι αν δεν έχουμε ευρωπαϊκή ενιαία αγορά θα πρέπει να εφεύρουμε μια ενιαία αγορά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι το οποίο υπονοεί κάποιες διατάξεις που θα ανταποκρίνονται στις διατάξεις κοινή αγοράς για το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχουν πει πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο, ούτε λέξη. Οπότε, αναμένουμε να δούμε το τι συνέπειες θα αυτό, γιατί δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά σε συγκεντρωτισμό. Η δεύτερη δυνατότητα είναι αντί για συγκεντρωτισμό το Ηνωμένο Βασιλείο να αποσυνδεθεί. Το έλεγε αυτό ο κόσμος πέρσι και πριν από έξι μήνες μετά το δημοψήφισμα. Βεβαίως λόγω των διαφορετικών αποτελεσμάτων μπορεί να διασπαστεί το Ηνωμένο Βασίλειο η Βόρεια Ιρλανδία να ενωθεί με την Δημοκρατία της Ιρλανδίας και η Σκοτία να κάνει ένα ακόμα δημοψήφισμα και να γίνει ανεξάρτητη για να παραμείνει εντός της Ένωσης. Και το επιχείρημα είναι ότι η Σκωτία ψήφισε να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά να παραμείνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα τους λένε «Ε, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να διαλέξετε μία από τις δύο ενώσεις. Οπότε η Σκοτσέζικη κυβέρνηση πρότεινε ένα ακόμα δημοψήφισμα. Το πρόβλημα εδώ είναι διπλό. Αφενός για να γίνει δημοψήφισμα χρειάζονται την έγκριση του Κοινοβουλίου του Westminster και δεύτερον, εάν γίνει ανεξάρτητη σκοτία εντός της Ένωσης θα έχουμε ένα σκληρό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ Σκοτίας και Αγγλίας όπως και στη Βόρεια και κανείς δεν το θέλει αυτό. Και συγκεκριμένα στην περίπτωση της Βορειοϊρλανδίας ε, έχουμε το σκληρό σύνορο όπω λέγεται και εν πάση περιπτώσει οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι από το δημοψήφισμα του 2014 δεν έχει αλλάξει η στήριξη της ανεξαρτησίας της Σκωτία. είναι ένα 45% συν 3. Εκεί είναι τα πράγματα, δεν έχει αναπηδήσει λόγω Brexit. Το τρίτον, σενάριο είναι η διαφοροποίηση. Σβήνει το μικρόφωνο του μιλτή. Α, κάτι θέλει να μου πει το μικρόφωνο. Μάλιστα. Θα μπορούσαν λοιπόν να βρουν την θέση τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της Ουαλίας βεβαίως δεν ασχολείται με αυτό, γιατί ε, ε, η Ουαλία δεν ψήφισε να φύγει, αλλά η κυβέρνηση της Σκοτίας ε, αναζητεί κάποιες προτάσεις, πώς μπορεί να παραμείνει εντός ενιαίας αγοράς η Σκοτία μόνο κτλ. Είναι περίπλοκα αυτά, τώρα δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι δεν είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί τέτοια ρύθμιση, αν και θα το κάνει για την Βορεια αλλά δεν είναι διατεθειμένο να το κάνει ε, για τη Σκωτία. Είμαστε λοιπόν σε δύσκολη θέση γιατί κανένα από αυτά τα τρία σενάρια δεν επιλύει τα προβλήματα. Τέλος, όσον αφορά τη Σκωτία και την Ουαλία, υπάρχει το θέμα του ρόλου τους στις διαπραγματεύσεις ε, της απόσυρσης. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι θα έχουν ένα βρετανικό Brexit, δηλαδή ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο θα ε, είναι στην διαδικασία. Υπάρχει μια μεικτή ε, Υπουργική Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις ε, που υποτίθεται ότι θα εισφέρει την άποψη των αποκεντρωμένων διοικήσεων στο Brexit. Βεβαίως συνεδριάζει σε άτακτα χρονικά διαστήματα. Δεν έχει συνεδριάσει από τις εκλογές, αλλά θα συνεδριάσει προσεχώς. Το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι οι κυβερνήσεις Σκοτίας και Ουαλίας έχουν πει ότι δεν είναι ικανοποιημένες με τον ρόλο τους στην διαδικασία γιατί θεωρούν ότι δεν τους στέλνουν τα έγγραφα εγκαίρως. Δεν μπορούν να παρέμβουν πριν το Ηνωμένο Βασίλειο συντάξει τα διάφορα έγγραφα και δεν ε, είναι στον μηνιαίο κύκλο των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν μεταξύ των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της κεντρικής κυβέρνησης. Το άλλο θέμα είναι το Γιβραλτάρ που είναι αρκετά διαφορετικό και καλό θα ήταν να μην αναμειγνύεται με την ε, αποκέντρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Είναι μια κτήση ε, του στέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και εμπίπτει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ε, εν περιπτώσει, επειδή έχει σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κι αλλιώ, συμμετέχει στην εσωτερική αγορά, αλλά όχι στην Τελωνιακή Ένωση, εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο ε, εδώ ε, με την νο, νότιο-ανατολική Αγγλία είναι η ίδια επικράτεια και ψήφισε στο δημοψήφισμα ε, ποσοστό 96% υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου ομόφωνη ήταν η ε, απόφαση να παραμείνουν. Αλλά βεβαίως πραγματικά ε, αφορά το Brexit και το Γιβραλτάρ ε, και δεν θα διατηρήσει τη θέση που θα έχει ε, ακριβώς επειδή είναι μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει αυτά να γίνονται μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά τα προβλήματα του Gibraltar δεν είναι τόσο περίπλοκα όσο της Σκοτίας και της Ουαλίας. Ε, το βασικό ζήτημα είναι η ελεύθερη κυκλοφορία και τα σύνορα. Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στις ε, ευρωπαϊκές και βρετανικές χρήματα αγορές ε, και ε, οικονομικές υπηρεσίες, αλλά το ουσιαστικότερο είναι ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο Γιβραλτάρ περνούν τα σύνορα και έρχονται από την Ισπανία κάθε μέρα, κυρίως είναι Ισπανοί και πολίτες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θέμα. Το Γιβραλτάρ θέλει τώρα να διατηρηθούν ανοιχτά τα σύνορα. Τεχνικά, κατά την άποψή μου, αυτό δεν ε, προκαλεί τεράστια προβλήματα. Κατά τα άλλα και η ε, η σκοτική κυβέρνηση είναι υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε σήμερα ελέγχους. Ενώ ε, στο Γιβραλτά υπάρχουν έλεγχοι. Ε, και εδώ υπάρχει ένα άλλο ενεχόμενο μέρος που είναι η Ισπανία. Και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει ε, η Ισπανία να εγκρίνει οτιδήποτε αφορά το Γιβραλτάρ ή τα. Άρα είναι τρία τα μέρη εδώ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Και αν μπορεί να βρεθεί μια συμφωνία με την Ισπανία, νομίζω ότι αυτά τα σύνορα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική και την πολιτική βούληση, αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν εμπόδια από πλευράς Βρετανικής κυβέρνησης για να χορηγούν διάφορες εξαιρέσεις στο Γιβρατάρ, ακριβώς επειδή δεν είναι τμήμα ε, ουσιαστικό του Ηνωμένου Βασίλειου όπως η, η όπως η ε, Σκοτία και η Ουαλία. Ευχαριστώ πολύ, καθηγητά Κίτιν. Έχουμε τώρα αρκετό χρόνο για ερωτήσεις, σχόλια. Η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε εξαιρετικές και πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο παρεμβάσεις. Πρέπει να σας πω καταρχάς ότι εγώ είμαι ευρωσκεπτικίστρια και ε, να πω το εξής. Υποθέτω ότι εσείς και οι δύο είστε υπέρ της παραμονής δεδομένου του ε, πανεπιστημιακού σας ε, ιστορικού και της κομματικής σας προτίμησης. Καλό είναι όταν έρχονται ε, διάφοροι ομιλητέ εδώ στα εργαστήρια να δηλώνουν και ε, πού ανήκουν. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα όσα είπατε, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν δύο-τρία σημεία που θα ενδιέφεραν το εργαστήριο να δούμε ποια είναι η θέση της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που εσείς λέτε. Και θα ήταν δίκαιο ε, να προβληθεί και αυτό. Και μπορείτε να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ, τι πρόσβαση έχετε σε στοιχεία της κυβέρνησης, της αυτής μεγαλειότητος. Έχετε ενημέρωση. Και ποια είναι η προστιθέμενη αξία τέτοιων εργαστηρίων. Και αυτά που μας παρουσιάσατε ε, για τις διάφορες αρχές και τους ορισμούς μπορούμε να τα αντιβαραβάλουμε με αυτά που θα μας πούνε εκπρόσωποι της ε, Βρετανικής κυβέρνησης της ε, Εγώ θεωρώ ότι πρώτα ότι είμαι Αγγλίδα και μετά Βρετανή. Και άκουσα ε, πρόσφατα κάποιο πολιτικό και ξέχοντα να λέει ότι όποιος δηλώνει Άγγλος τις τελευταίες μέρες ε, θεωρείται ρατσιστής. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα. Ε, κατά τα άλλα έχω και σκοτσέζικο αίμα, αλλά θεωρώ ότι είμαι Αγγλίδα γιατί γεννήθηκα στην Αγγλία. Οι Σκοτσέζοι είναι πάρα πολύ περήφανοι όταν δηλώνουν Σκοτσέζοι. Άρα ο κόσμος δεν θέλετε να είναι προσιλωμένος στην πατρίδα του και με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Εντάξει, ε, για την ιστορία, πώς δημιουργήθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο. Και με πολέμους και με εισβολή αν θέλετε και με επιθέσεις, αλλά υπήρχε και πάρα πολύ εθελούσια ένωση ε, λόγω της δινής οικονομικής θέσης στην οποία βρισκόταν η Σκοτία, ε, οπότε συμφώνησε να μοιραστεί την εξουσία και την κυριαρχία με το Westminster. Παρακαλώ αυτά που μας εξηγείτε μπορείτε να τα τσεκάρετε κιόλας. Και ένα τελευταίο αναφερθήκατε ε, για το νομοσχέδιο για την ανάκληση της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας, the Great Repeal Bill. Εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο και εγκριθούν όλοι οι νόμοι και περάσουν από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, Αυτό σας καθησυχάζει ή όχι. Γιατί έχουν αποθέσει πολλές ελπίδες σε αυτό το νομοσχέδιο για την προστασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αν εσείς κατά κάποιο τρόπο ε, ισχυρίζεστε ότι δεν λαμβάνετε υπόψη, θα ε, μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τις απόψεις σας. Και ένα τελευταίο, ε, ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ. Το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκοτίας θα πρέπει να ε, εξετάζεται τελείως χωριστά από ε, το ε, δημοψήφισμα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι που λέτε ότι δεν είναι δεσμευτικό. Και αν έχει την ευκαιρία τώρα η Σκωτία να ξανακάνει τέτοιο δημοψήφισμα, να σας θυμίσω ότι οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Σκοτσέζοι δεν θέλουν δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία σε ποσοστό 60%. Ευχαριστώ πολύ. Η Ε, Ευχαριστώ, παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας. Ευχαριστώ. Που αυξήσατε το επίπεδο της περιπλοκότητας της καταστάσεως. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις δύο παρεμβάσεις. Είπατε ότι τα σύνορα θα πρέπει, με σειρά τα λέω, θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορα στην Ιρλανδία, μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ιρλανδίας, να μείνουν ανοιχτά μεταξύ Σκοτίας και ενδεχομένω Ουαλίας με την υπόλοιπη Ευρώπη και στο Γιβραλτάρ. Το μόνο σημείο που πρέπει να υπάρξει σύνορο θα ήταν μεταξύ Ουαλίας και Βρετανίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι. Μεταξύ Ουαλίας και Αγγλίας μάλλον, συγχωρείτε. Από όλα αυτά που είπατε αυτό καταλαβαίνω. Έτσι λύνεται και το πρόβλημα της Βορείου Ιρλανδίας. Διότι τα σύνορα με την Αγγλία, με την Ουαλία θα ήταν τα μόνα που θα έμεναν. Είναι ένα παράδοξο θα έλεγα αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να εκφράσω κάποιες ανησυχίες που άκουσα. Πολύ πιο δύσκολο φαίνεται το θέμα του σκληρού Brexit. Αν η επιλογή είναι το soft Brexit, δηλαδή να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην ενιαία αγορά και στην Τελωνιακή Ένωση, είναι ξεκάθαρο ότι βασικά προβλήματα επιλύονται, εκτός από κάποια που αφορούν τους ευρωπαϊ... τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τη γεωργία ή για άλλες δραστηριότητες. Αναπτυξιακή πολιτική, Φερρυπίν. Για Σκοτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία. Όμως αυτά μπορούν να επιληθούν δεν θα πληρώνει πλέον συνεισφορές το Ηνωμένο Βασίλειο και θα κάνει δική του πολιτική για τη στήριξη της Γεωργίας. Εκεί που θα πρέπει να δίδεται για τη συμμετοχή στην ενία αγορά. Θα ασκήσει πολιτική εσωτερική συνοχής. Δεν μπορεί να τον εμποδίσει, να εμποδίσει κανείς το Ηνωμένο Βασίλειο να το κάνει αυτό. Είναι εσωτερικό θέμα. Δεν κατανοώ Μια άλλη λύση που να μπορεί να δώσει απάντηση σε όλα τα προβλήματα που υπογραμμίσατε. Είναι προφανέστατο ότι το πρόβλημα ελέγχου των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι κάτι που έχουμε ακόμα πρόσφατα. Συζητούνται πάμπολα προβλήματα που έχουμε. Τελωνιακά ήδη υπάρχουν με το Ηνωμένο Βασίλειο Υπάρχει διαδικασία επί παραβάση. Εν γέννη θα ήταν πολύ δύσκολο να δεχτούμε ρευστά σύνορα, ανύπαρκτα σύνορα ή πολύ μαλακά ούτως υπήν σύνορα. Ερώτηση. Κατά την άποψή σας, μπορούμε να εξετάσουμε περισσότερο ένα μοντέλο που το ξέρω προσωπικά, που ισχύει με την Ελβετία. Η Ελβετία ανήκει εν μέρη στην ενή αγορά. Δεν ανήκει στην Τελωνιακή Ένωση. Σε αντιστάθμιση όμως ανήκει στο Σέγγεν. Και υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία. Η έλεγχοι γίνονται στα εμπορεύματα. Όχι σε ένα πακέτο, ένα δέμα μεταφέρει κάποιος, αλλά ελέγχονται τα μεγάλα φορτία στα σύνορα. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορούσε να εξεταστεί. Θα έλυνε το πρόβλημα ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων, βέβαια όχι των εμπορευμάτων. Αλλά το θέμα των εμπορευμάτων ρυθμίζεται πιο εύκολα. Άλλο ενδεχόμενο, που ίσως ανέφερε ο συνάδελφος Κόρμπετ στην περίπτωση Βορείου Ιρλανδίας τα σύνορα Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορούν να μετακινηθούν και να πάνε στα λιμάνια της Βορείου Ιρλανδίας και να τα χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε η Ιρλανδία να παραμείνει ελεύθερη όσον αφορά τις εσωτερικές μετακινήσεις, αλλά όχι ενάντια του εξωτερικού, διότι είναι δύσκολο αυτό να το επιτρέψει να γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια ερώτηση. Η κυρία Τσιούντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Childers. είμαι βουλευτής από την ε, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ανήκω στους σοσιαλιστές, είμαι ευρωβουλευτής. Απλή ερώτηση. Πώς το κρίνετε. Περιγράψατε πολύ περίπλοκα θέματα και τα επίπεδα περιπλοκότητας αυξάνονται καθημερινά. Βλέποντας δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διαθεσή μας Πώς θα λυθεί το θέμα. Και τελικά ίσως να καταρρεύσουν εντελώς οι διαπραγματεύσεις, γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκες. Όπως ο πρώην Υπουργός, ε, Οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης, περιέγραφε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν το, hotel, σαν το ξενοδοχείο Καλιφόρνια. Μπορούσε να μπει, αλλά δεν μπορούσε να βγει. Και δεν ήταν υπέρ του Brexit που εξέπληξε κάποιου. Δοθήσει τη καταστάσεω. ότι η δημοκρατία της Ιρλανδίας αντιμετωπίζει ενδεχομένω φρικτά προβλήματα. Είναι σε χάλια λόγω αυτού του ενδεχομένου. Ποιο είναι το λογικό χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταβατικό για την αποχώρηση. Πιθανότατα δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι το άρθρο 50 ποτέ δεν θεωρείται ότι θα ενεργοποιηθεί. Θεωρείται σαν αποτρεπτικό άρθρο. Αν Τρία χρόνια, εφτά χρόνια θα μπορούσε να είναι μια μεταβατική περίοδος μακρύτερη που θα επέτρεπε επίλυση προβλημάτων. Ποια είναι η άποψή σα. Ποιο χρονικό διάστημα θα διευκόλυνε κάπως αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Σε εσά το λόγο και μετά θα έχουμε άλλο ένα γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να απαντήσω στην Ταϊάν πρώτα. Πρώτα απ' όλα η θέση μου. Εγώ θα έλεγα ότι είμαι ένας αντικειμενικός ουδέτερος ε, πανεπιστημιακός. Το ωραιότερο πράγμα που μου έχουν πει ποτέ είναι μια φοιτήτρια μετά από τρία χρόνια μου είπε ακόμα δεν ξέρουμε πώς ε, ψηφίσατε και το ίδιο θα ήθελα να ισχύει για το δημοψήφισμα. Έχω μια θέση δεδομένου του ότι βεβαίω ο Πρίτανή μου ήταν υπέρ της ε, παραμονής θα ήταν κάπω ίσως όχι έξυπνο να είμαι υπέρ του Brexit αλλά τέλος πάντων θα έλεγα ότι το έγγραφο της ε, κυβέρνησης ε, για την Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία ήταν μεγάλη πρόοδος σε σχέση με την ε, Λευκή Βίβλο των αρχών του 2017 που έμοιαζε ένα συμπίλημα κάπως και δεν είχε σχοληθεί καθόλου με το θέμα της Βόρειου Ιρλανδίας. Εν ήταν κάτι το χρήσιμο ε, επαναλάμβανε το πού βρίσκεται η κυβέρνηση και βεβαίως ο βασικός στόχος ήταν να υπάρχει ένας κοινός ταξιδιωτικός χώρος, κάτι το οποίο είναι βεβαίως πάρα πολύ καλό. Ε, υπάρχουν βεβαίως ε, κάποιοι λόγοι μεταναστευτικής πολιτικής της Βρετανίας, δηλαδή αν θέλει να μπει κανείς από το παράθυρο πάει στην Ιρλανδία, τη δημοκρατία γιατί δεν θα υπάρχει έλεγχος σε εκείνο το σύνολο. αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα στην Ιρλανδία. Δεν ήταν αυτό το κίνητρο στην Βόρεια Ιρλανδία. Το θέμα εκεί ήταν η ταυτότητα, αν αισθανόταν περισσότερο ή Ιρλανδή Και δεν αφορούσε ούτε την κοινωνική τάξη, ούτε την ηλικία. Οπότε όλα αυτά που ακούσαμε για το δημοσίευμα στην Αγγλία, Σκοτία και η δεν ισχύουν για την Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε θα μπορούσε να υπάρχει ένας κοινό ε, χώρος ε, για την μετακίνηση και ο David Davis ήταν σαφέ ότι δεν θα υπάρχουν κάποια φυσικά εμπόδια στα σύνορα και βεβαίω αυτό συμφωνεί και με την Ιρλανδική κυβέρνηση. Το θέμα είναι όμω αν επιτρέπεται κάτι τέτοιο και νομίζω ως ένα βαθμό ε, έχει επιστρέψει το μπαλάκι στην Ιρλανδική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Τώρα, εκεί όπου είναι αμφίσιμη η Βρετανική θέση είναι το σε ποιο βαθμό έχει αποκλείσει την πρόσβαση στην Τελωνιακή Ένωση. Έχει πει ότι δεν θα είναι μέρος της Τελωνιακής Ένωσης γιατί είναι θέμα κυριαρχίας και εμπορικών συμφωνιών με άλλους, αλλά είναι ακόμα σαφές για το εάν είναι διατεθειμένη να πληρώσει για πρόσβαση στην Τελωνιακή Ένωση. εάν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο, για να λυθεί το πρόβλημα του σύνορου στην ίσο της Ιρλανδίας και όσον αφορά τα δεδομένα της κυβερνήσεως της αυτής ε, μεγαλειότητος. είχα καταθέσει και στην Βουλή των Λόρδων, στην ανάλογη επιτροπή και χρησιμοποίησα δικά τους δεδομένα, έκαναν πολύ καλές εκθέσεις και κυρίως αυτά τα δεδομένα έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και ο Νταν Τζέιμς ε, έχει δίκαιο, δεν θα πω πώς ψήφισα σε αυτό το δημοψήφισμα όπως και στο σκοτσέζικο δημοψήφισμα και σε οτιδήποτε άλλο είναι ζήτημα νομίζω και επαγγελματική διοντολογίας. Είμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, με τα διάφορα υπουργεία και με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Έχουμε ελεύθερη πρόσβαση και για ενημερώσεις soft record και για δημόσιες ενημερώσεις και νομίζω ότι όλες οι πλευρές το θεωρούν αυτό επικοδομητικό γιατί βεβαίω είμαστε και διακριτικοί και υπάρχει κάποια ηχεμήθεια. Το άλλο, α, δεν το ανέφερα, πώς ε, βλέπουμε την Αγγλία γιατί πραγματικά αμελείται εντός του συντάγματος αλλά αυτό δεν ήταν ε, τμήμα της ε, Λοιπόν, πράγματι είναι μια εθελοντική ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό έλεγα. Και συνεχώς τα έθνη διαπραγματεύονται την θέση τους εντός αυτής της ένωσης. Και βεβαίω αυτό σημαίνει και συνένεση των άλλων εθνών. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 20 χρόνια και δυσκολεύει λόγω του Brexit για την νομοθεσία περί απόσυρσης του, κατάργησης του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, ασχολείται με ακριβώ αυτές τις αλληλεπικαλύψεις ε, αρμοδιοτήτων που υπάρχουν, που θα επανέλθουν στο Westminster και εκεί πέρα θα αποφασίσει το Westminster τι θα πάει στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Βεβαίω εδώ πέρα ανησυχούν ιδιαίτερως οι κυβερνήσεις Σκοτίας και Βαλίας και έχω σχολιάσει και στο blog μου και αλλού πως υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα γιατί βεβαίως ε, εδώ πέρα καθορίζουμε τις ε, αρμοδιότητες ε, με βάση το τι έχει νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το τι είναι όντως αρμοδιότητα και αυτό φοβάμαι ότι θα μας απασχολεί στα δικαστήρια στο μέλλον. Κύριε Μπρέσο λέει για τα σύνορα όλοι θέλουν να ανοιχτά σύνορα. Ναι, ναι, αυτή είναι η αρχική θέση όλων και είναι πολύ σημαντικό, αλλά το ερώτημα είναι πώς κάνουμε κάτι τέτοιο και το Brexit και η αποκέντρωση ακριβώς ε, αφορούν και τα μεταβαλλόμενα σύνορα. Να τα σεβόμαστε, αλλά να γίνουν και πιο διαπερατά. Ε, ακόμα και αν υφίστανται. Το θέμα ενός ήπιου Brexit, ναι, αυτή είναι η προτίμηση της κυβέρνησης της και η δεύτερη, η τρίτη θα έλεγα προτίμηση της σκοτίας. Δηλαδή αν δεν λάβουν αυτό το οποίο θέλουν θα προτιμούσαν να είπε ο Brexit γιατί η Σκοτία και η Ουαλία θα ήθελαν την εσωτερική αγορά και ίσως και την Τελωνιακή Ένωση και ειδικά η Σκοτία είναι υπέρ της ελεύθερης μετακίνησης ε, και να είπε ο Brexit θα έλυνε πολλά από αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό και οι δύο κυβερνήσεις πηγαίνουν προς τον... υποστηρίξουν τον συνασπισμό του ήπιου Brexit που είναι μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου και του Συντηρητικού Κόμματος και ίσως το μισό εργατικό κόμμα και τους ε, φιλελεύθερους δημοκράτες και τους πράσινους. Είναι βλέπετε το ζήτημα οριζόντιο και τέμνη τα κόμματα. Οπότε εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα πάμε σε Brexit και έτσι, αυστηρά σύνορα. Το ελβετικό μοντέλο έχει αναφερθεί, αλλά η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει το ελβετικό μοντέλο γιατί είναι περίπλοκο. Υπάρχουν 120 διμερείς συνθήκες. Υπάρχει βεβαίως ελευθερία μετακίνηση και ακριβώς αυτό προκάλεσε πρόβλημα στους Ελβετούς πριν από δύο χρόνια και λέει δεν θα το δεχτεί η Δεθνική Κυβέρνηση. Τώρα για την Ιρλανδία και το σύνορο το Βρετανο-Ιρλανδικό θα, είναι μια, ε, θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά βεβαίως ε, οι ενωτικοί στην Βόρεια δεν θα το δεχόντουσαν. Για την μεταβατική περίοδο δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, γιατί υπάρχει όντως μια αμφισημία. Τι σημαίνει, ότι θα κάνουμε όλες τις διαπραγματεύσεις, θα ξέρουμε το πού θα καταλήξουμε το Μάρτιο του 2019 και μετά θα το εφαρμόσουμε ή συνεχίζομαι, ή συνεχίζονται, με συγχωρείτε οι διαπραγματεύσει σε όλη αυτή την περίοδο. Δεν είναι σαφή και δεν ξέρω και τι εννοεί η κυβέρνηση. Η Βρετανική, το τελευταίο αυτό βεβαίω δεν μπορεί να γίνει, αλλά αυτό φαίνεται ότι προτείνει η κυβέρνηση ότι η τελική συμφωνία θα προκύψει κατά τη διάρκεια τη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφεί. Η Τερίζα Μέη μιλάει για περίοδο εφαρμογή, οι άλλοι λένε μεταβατική περίοδο. Αυτό το οποίο είναι σαφέ είναι ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια. Όλοι συμφωνούν. Κάποια πράγματα απλά θα τα αφήσουμε κατά μέρο ή θα τα αφήσουμε όσο έχουν. Και δεν ξέρουμε πώ θα γίνει κάτι τέτοιο. Κάποιε από τι προσωρινέ αυτέ διευθετήσει, ίσω τελικά μα συνοδεύσουν για καιρό. Ε, σύντομα, συμφωνώ με τον Μάικλ για το ελβετικό μοντέλο. Είναι πολύ περιπλοκό. Ίσως για κάποιου τομεί θα μπορούσε να ισχύσει π.χ. για το εμπόριο μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Ιρλανδικής Δημοκρατίας. Αλλά για το πού ε, θα ήταν το σύνολο. Εκεί πέρα οι ενωτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία επιμένουν ότι δεν θέλουν έλεγχο διαβατηρίων από το ένα κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου στο άλλο, για να πάνε δηλαδή από τη Βόρεια Ιρλανδία στο Λίβερπουλ ή στη Σκωτία. Είναι κόκκινη γραμμή για τους ενωτικούς του Άλστερ ότι δεν είναι διατεθειμένοι να τους ελέγχουν τα σύνορα. Θεωρούν ότι είναι μέρος του ε, Ηνωμένου Βασιλείου. Βεβαίω οι Ιρλανδοί εθνικιστέ έχουν διαφορετική άποψη. Ε, αυτό το οποίο είπατε. Ναι, δηλαδή μετάβαση σε τι. Μέχρι στιγμή η Βρετανική κυβέρνηση απλά χρονοτριβεί. Δεν μπορεί τέτοιε εμπορικέ συμφωνίες να συναυθούν σε δύο χρόνια. Δηλαδή μετάβαση σε μια συμφωνία του ΠΟΕ. Αυτό χρειάζεται να δύο χρόνια. Εγώ έτσι το βλέπω αυτή τη στιγμή. Thank you. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος δίνει το λόγο στον κύριο Κόρμπετ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι ήταν εξαιρετικές οι παρουσιάσεις. Έθεσαν τα προβλήματα και τα διλήμματα που απορρέουν από το Brexit. Πρέπει να ομολογήσω ότι απογοητεύτηκα πολύ από την ερώτηση που σας έκανε η κυρία Τζέιμς. Και στόχο είχαν να σας βάλουν ταμπέλες και να προσπαθήσουν να ε, σας κατατάξει κάπου, να πει ότι μεροληπτείτε και να αφαιρέσει την αξιοπιστία των λεγόμενων σας. Μα τίθενται ζητήματα τα οποία κανείς δεν έθεσε και κανείς δεν συζήτησε, ούτε εξήγησε σε λεπτομέρειες κατά το δημοψήφισμα και όλα αυτά αναδεικνύονται και καταδεικνύονται από τα όσα λέτε. Και το γεγονός ότι είναι πρόθυμη η κυρία Τζέβης να δώσει αυτή τη μάχη δείχνει ότι δεν έχει χωνέψει ο κόσμος ότι έχει λήξει το Brexit και ότι πρέπει ακόμα να αγωνίζεται σε αυτό το πεδίο. Χαίρομαι που λέτε και να γνωρίζετε ότι υπάρχει ακόμα ε, αντιπαράθεση ως προς το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να έρθω στην ερώτησή μου τώρα για τα σύνορα Βορείου Ιρλανδίας και ε, Ιρλανδικής Δημοκρατίας. Αναφέρετε διάφορες ε, δυνατότητες και διάφορα προβλήματα που συνδέονται με την κάθε μία εκδοχή η μόνη πολιτικά βιώσιμη λύση και τεχνικά και τεχνολογικά εφικτή, αν υποθέσουμε ότι θα αποχωρήσει η ε, Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να παραμείνει στην Τελωνιακή ε, Ένωση Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Put the microphone Ο κύριος Γκίλ. Ε, κύριε καθηγητά Κίτσινγκ, περιγράψατε το Γιβραλτάρ ως μια κτήση του στέματος, crown dependency. Δεν είναι αρ, ε, ακριβές αυτό. Είναι μια υπερπόντια κτήση με δική της βουλή, σύγχρονο σύνταγμα και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μόνο αρμόδιο για την εξωτερική και εσωτερική του ασφάλεια. είχα την ευκαιρία να μεταβώ εκεί και να δω ε, με πόσο ρεαλισμό αντιμετωπίζουν το Brexit. 96% ψήφισε υπέρ της παραμονής. Εγώ που είμαι οπαδός του Brexit προβληματίστηκα Πώς είναι δυνατόν μια επικράτεια που αυτοχαρακτηρίζεται βρετανική και είναι πάρα πολλοί πατριώτες, πολύ περισσότερο από τους υπολείπους του Ηνωμένου Βασιλείου, αποφάσισαν να παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πήγα εκεί και είδα ότι το μεγαλύτερο κίνητρό τους ήταν ο φόβος ε, ως προς το τι θα γίνει με τα σύνορα. Και τι αποφάσισαν λοιπόν. Θεώρησαν και προεξόφλησαν ότι το Brexit είναι πραγματικότητα και επειδή είναι ρεαλιστές αποφάσισαν το καλύτερο που έχουν να κάνουν να δουν τις επιπτώσεις και το, πώς θα πετύχει το Brexit για το Γιβραλτάρ. Και αντί να χρονοτριβούν και να προσπαθούν να ε, το παρουσιάσουν ωραιοποιημένο, ήπιο το Brexit, νερόβραστο κτλ. Ε, ε, λένε ότι, ωραία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς πιστεύουμε στην ενιαία αγορά, το 90% του εμπορίου τους είναι με το Ηνωμένο Βασίλειο, το υπόλοιπο 10% με την υπόλοιπη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, είναι εκτός της Ελληνικής Ένωσης ήδη και έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο, είναι ρεαλιστές, ε, ευτυχισμένοι, αισιόδοξη, στραμμένη προς το μέλλον. Και αυτό είναι και ένα δίδαγμα για όλους στο Ηνωμένο Βασίλειο που ζουν σε περιοχές που ψήφισαν υπέρ της παραμονής. Ε, και τώρα πρέπει να το δεχτώ. Εγώ είμαι από την Ολία. Έχουμε τέσσερι ευρωβουλευτέ από την Ολία. Η Ολία ψήφισε υπέρ του Brexit. Τώρα θα πρέπει να δεχθούμε ε, ε, την λαϊκή ετοιμιγορία. Σταματείτε να επανα προσδιορίζεται να επανορίζεται το Brexit. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε, όπως το Γιβραλτά. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε όλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον ίδιο ρεαλισμό. Okay, then I... Ευχαριστώ πολύ. Να θέσω εγώ ερώτηση. Ουδής άλλος επιθυμεί. Θεωρητικό ερώτημα. Σας αρέσει κιόλα. Mm. καθηγητής Κίτη αναφέρθηκε στο Σύνταγμα. Λειτουργούν οι συνελεύσεις για το Σύνταγμα μόνο αν υπάρχει μια νοοτροπία αυτοπεριορισμού που επικρατεί. Κάτι που απέδειξε ιστορικά η χώρα. Άρα, η έλεγχη είναι πολύ αποδυναμωμένη στον Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε στην κυριαρχία του Westminster, της Βουλής των Κοινοτήτων, που δεν ελέγχεται. Αυτές αυτά τα θέματα δεν λύνονται εύκολα όσον αφορά την ταυτότητα. Και ιδίω με κάποιο τρόπο είπατε ότι κάποια από τα στοιχεία χαρακτηρίζονται από την έννοια της ταυτότητας. Ρίχνω την ερώτηση. Χρειάζεται συνταγματική συνέλευση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να ετοιμαστεί ένα πραγματικό σύνταγμα σαν αυτό που έχουμε εμείς από την άλλη πλευρά της μάχης. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα χωρίς εκ νέου τοποθέτηση πλαισίου, εγώ διαβλέπω συνεχή τριβή μετά το Brexit όταν πραγματοποιηθεί, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα πραγματοποιηθεί. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Ε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Σαφέστατη ερώτηση. Αν μόνη λύση είναι να μείνουμε στην Τελωνιακή Ένωση η πιο ελκυστική είναι θα έλεγα υπό διάφορους όρους. Από πολιτική σκοπιά θα πρέπει το Ενωμένο Βασίλειο στο σύνολό του να παραμείνει στην Τελωνιακή Ένωση. Λόγω αντιρρήσεων των ενωτικών για το ειδικό καθεστώς για τη Βόρεια Ελλανδία και να παραμείνει στην ε, Τελωνιακή Ένωση. Θα δοθεί ένα επίπεδο αυτονομίας στη Βόρεια Ελλανδία που δεν είδαμε προηγουμένως εκτός από τη δεκαετία του 70 που είχαν εκχωρηθεί ε, δικαιώματα και αυτονομία. Θα ήταν δύναμή τη τέτοια αυτονομία. Θα πρέπει να ισχύσει για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπαίνουμε σε πιο βαθιά νερά μετά. Βλέπουμε το τουρκικό μοντέλο τη Θελωνιακή Ένωση που παρατίθεται συχνά, σαν παράδειγμα. Ποιο είναι το πρόβλημα όσον αφορά μοντέλο. Δεν καλύπτει τη Γεωργία, και θα ήταν γελίο κάτι τέτοιο για τη Βόρεια Ιρλανδία που είναι βασικό εξαγωγικό προϊόν του γεωργικού τομέα. Μπορείτε να έχετε τελωνιακή συμφωνία που καλύπτει όλους τους τομείς. Αυτό ξεπερνιέται. Μετά υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυριαρχία την εμπορική του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν η Εάν δεν μπορούν οι συμφωνίε τη Ελληνική Ένωση να επιτρέψουν σε συμβαλόμενα κράτη να συνάψουν συμφωνίε διμερεί με άλλα κράτη, είναι πρόβλημα. Αυτοί που υπερασπιζόταν ε, το Brexit ήθελαν και αυτό. Και γι' αυτό θέλαν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η Βρετανική κυβέρνηση δεν ήθελε να δεσμευτεί να παραμείνει στην ε, Τελωνιακή Ένωση, αλλά έδωσε τη λύση πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι με Τελωνιακή Ένωση στα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα πληρώνονται πολλά χρήματα στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτρέπεται το εμπόριο χωρί δασμού κλπ για να λυθεί το πρόβλημα των συνόρων στην ίσο της Ιρλανδίας. Αυτό είναι εφικτό. Μπορεί να το πωλήσει κανείς και στις δύο πλευρές, και σε αυτούς υπέρ του Brexit και σε αυτούς που είναι κατά. Αλλά πρέπει να είναι κομμένο και ραμμένο, κομμένη και ραμμένη συμφωνία στα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Γίνεται, ενδεχομένω. Αλλά σωστή η βασική υπόθεση της ερώτησής σας. Ίσως είναι η μόνη επιλογή για να αντιμετωπιστεί το θέμα των συνόρων στην ίσο της Ιρλανδίας. Αλλιώς θα πρέπει να επιβληθεί κάποιο τελωνιακό καθεστώς. Τώρα συνταγματική συνέλευση. Ναι, αλλά σε ποιο βαθμό θα διευθετήσει τα αναφερθέντα προβλήματα. Εγώ θα πρότεινα κάτι κάτι σαν συνέλευση των πολιτών, όπως στην Ιρλανδία, που έκανε διάφορες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και εγώ πρέπει να πω ότι το έβλεπα θετικά, αρχικά. Άρα καλύτερες προτάσεις και πιο δημοκρατικές προτάσεις βγαίνουν από κάτι τέτοιο. Παρά να κάνει προτάσεις ε, μια ελίτ μέσω συντακτικής συνελεύσεως. Ίσως το μοντέλο αυτό που ακολουθήθηκε στην Ιρλανδία να ήταν καλύτερο. Για την ερώτηση για το θέμα του Γιβραλτάρ. Λιγότερα και τα προβλήματα σε σχέση με τις, ε, με τις αποκεντρωμένες εξουσίες του ΕΒ. Δεν ανήκει στο ΕΒ το Γιβραλτάρ. Έχει τις αρμοδιότητες να αντιμετωπίσει τα θέματα του Brexit ήδη διαφορετική θέση του έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκρίση με οτιδήποτε τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θεωρώ ότι δημιουργεί προηγούμενο. Έχει τι εξουσίε που ζητούν ε, η Ουαλία και η Σκοτία. Έχει δική του διμερή ε, Διπουργική Επιτροπή με το Ηνωμένο Βασίλειο και θα λυθεί το θέμα μεταξύ Ισπανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, χω, χωρίς να υπάρχει σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη Σκωτία. Τώρα, τι γίνεται με τα σύνορα στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό έχω να πω. Όσον αφορά τι συντακτικέ συνελεύσει. Ναι, σωστά το είπατε. Λειτουργούν αν υπάρχει αυτός, αυτή η νοοτροπία του αυτοπεριορισμού. Και αν αυτό καταρρεύσει, συντάσσουμε γραπτό σύνταγμα. Και όταν υπάρξει με τέτοια κρίση, να πλησιάζουμε τέτοια κρίση τώρα μπορεί να επιληθεί με συντακτική συνέλευση. Είμαι πολύ διστακτικός. Αυτοί που προτείνουν συντακτική συνέλευση λένε ότι αφορά όλα αυτά επί των οποίων συμφωνούμε. Επί των περισσότερων θεμελιωδών ζητημάτων, κράτος δικαίου, ε, δημοκρατία κλπ. Ε, συμφωνούμε. Ποια θα είναι η φύση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πολυεθνική ένωση, ε, ενιαίο κράτος κλπ. Και μπορέσαμε να αποφύγουμε αυτό το θέμα, το αφήσαμε κάπου παράμερα. Δεν συμφων... Εάν δεν συμφωνούμε είπαμε γιατί να το κουβεντιάζουμε. Απλώς φάβουμε ε, τις διαφωνίες. Αν οι δύο πλευρές στη Βόρεια Ιρλανδία δεν μπορούν να συμφωνήσουν και να καθίσουν σε τραπέζι κάπου αλλού στο νησί και να συμφωνήσουν και οι... με τους Σκοτσέζους και οι Σκοτσέζοι με τους Άγγλους, πώς θα γίνει αυτό στο μέλλον ίσως αλλάξουν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί κάτι Είναι πολύ ρευστή η περίοδος. Είναι τόσο μεγάλη η ρευστότητα που οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι πάρα πολύ προσωρινή. Τώρα δεν είναι στιγμή για κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό στη διαδικασία του Brexit. Θα είναι υπερφόρτωση. Εν τη διαδικασία του Brexit, ίσω δημιουργηθούν πολλά προηγούμενα που θα δεσμεύσουν και το μέλλον. Αυτή τη δυσκολία αντιμετωπίζουν. Προχωρούν πολύ γρήγορα τα πράγματα και αλλάζει το Σύνταγμα μπροστά στα μάτια μα. Πολύ συχνά χωρί να κατανοούμε ποια είναι η κατεύθυνση και τι κάνουμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε κατανοητό στον κόσμο ποιε είναι οι γενικότερε συνέπειε. Οι βραχυπρόθεσμε, όχι οι μακροπρόθεσμε τόσο αλλά έχουμε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας. Περισσότερες συνταγματικές αλλαγές που είχαμε τα τελευταία 100 χρόνια γίνονται τώρα. Ευχαριστώ, πολύ. Ο Ραμόν Χάουρεκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είχα την πρόθεση να ζητήσω το λόγο. Pero ha surgido... Αλλά επειδή ανέκυψε το θέμα του Γιβραλτάρ, συμφωνώ απολύτως ε, με αυτά που λέτε. Ε, ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ε, μεταξύ των περιπτώσεων που συζητούμε. Άλλο Ηνωμένο Βασίλειο, Σκοτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και άλλο Γιβραλτάρ. Ωστόσο, με εξέπληξε η υπεραισιοδοξία του συναδέλφου μου ε, για το βρετανικό πατριωτισμό στο Γιβραλτάρ που θα οδηγήσει τον κόσμο σε μια θαυμάσια λύση στο περιθώριο της Ευρώπης δεν μπορώ παρά να σας εκφράσω την ανησυχία μου για το μέλλον των κατοίκων του Γιβραλτάρ υπό την έννοια αυτή. Γιατί ουσιαστικά και πραγματικά δεν πρόκειται μόνο για τα σύνορα τους, αλλά και για το εμπόριο, τη βιομηχανία που έχουν ε, εκεί του το, τζόγου, ε, ε, τα φορολογικά, όλα τα χρηματοπιστωτικά. Όλα αυτά σήμερα είναι συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σκεφτούμε ξαφνικά ότι μετά το Brexit θα έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν. 28.000 είναι οι κάτοικοι που βεβαίως έχουν 22.000 εταιρείε. Έτσι κάθε κάτοικος μία εταιρεία περίπου. Και θα έχουν τη δυνατότητα αυτή να χτίσουν το μέλλον τους στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μου φαίνεται πραγματικά ανησυχητική αισιοδοξία για εκείνους. Και επιτρέψτε μου να σας πω κυρίες και κύριοι ότι το Γιβραλτάρ και η Ισπανία θα πρέπει να συνεννοηθούν γιατί ζουν κολλημένοι. Ο ένας με τον 10.000 είναι οι Ισπανοί εργαζόμενοι που κάθε μέρα περνούν τα σύνορα για να εργαστούν και το βράδυ επιστρέφουν. Και δεν πρόκειται μόνο για τους εργαζομένους. Είναι ολόκληρο το πρόβλημα που έχει ο βράχος του Γιβραλτάρ. Ένα αέριος χώρος, λιμένας, ε, μεταφορές κλπ. Είναι ένα σύνολο προβλημάτων. Το μέλλον του Γιβραλτάρ θα πρέπει να εγγραφεί επίσης σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πέρα από τα ποσοστά του εμπορίου για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι τελείως ε, εξωπραγματικό να σκεφτόμαστε το μέλλον του Γιβραλτάρ σαν να μην υπάρχει η Ευρώπη. Η Ισπανία λοιπόν και το Γιβραλτάρ πρέπει να συνεννοηθούν και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εσείς θα πρέπει να καταλάβετε ότι η Ισπανία διατηρεί μια πολιτική αντίληψη για αυτό το χώρο. Εμείς το θεωρούμε απικία. Το έχει αναγνωρίσει και ο ΙΕ και ζητούν μια λύση να βρεθεί, το συστήνουν τα Ηνωμένα Έθνη ε, στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαπραγμάτευση είπε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν η Ισπανία και η Ηνωμένο Βασίλειο. Και δεν πρόκειται ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί καμία συμφωνία για το Γιβραλτάρ εφόσον δεν έχουν προηγουμένως συμφωνήσει η Ισπανία και η Ηνωμένο Βασίλειο. Τελεία. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Πάντως πρέπει κάτι να γίνει για να υπάρξει τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε. Χρόνο έχουμε. Κοιτάξτε, και εμένα δεν ανέφερα το θέμα Ισπανίας ε, Μεγάλη Βρετανία για το Ιβρυματάριο. Το γνωρίζω, αλλά δεν θα πω τίποτα. Να πω μόνο να επαναλάβω ότι το θέμα του Γιβραλτάρ ε, διαφέρει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ακριβώς να κάνει με τα σύνορα και νομίζω ότι αναγνωρίζουν όλοι ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οποιαδήποτε απόφαση για τα σύνορα θα πρέπει να εγκριθεί και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν αφορά μόνο τους Ισπανούς πολίτες, όπως στην Ιρλανδία, αλλά και τους άλλους ε, Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στην Ισπανία. Αλλά τεχνικά δεν βλέπω κάποιο εμπόδιο είναι θέμα πολιτικής βούλησης για να γίνει κάτι τέτοιο. Και οπωσδήποτε το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα παραμείνει, γιατί αυτή η διάσταση αφορά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ναι. ότι τελειώσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο καθηγητές. Είχαμε μια συναρπαστική ναι. συζήτηση. Εγώ έμαθα πολλά, πολύ διαφωτιστική. Επαναλαμβάνουμε τη συνεδρίαση στις 5. Ε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να συνταχθούμε λίγο. Πάντα ήθελα έτσι να έχω το σφυράκι μου. Okay, when? Ah, okay. Right. So, may we, may we come to order? Λοιπόν, ανασύνταξης παρακαλώ, για να επαναλάβουμε τη συνεδρίασή μας. Έχω να σας κάνω ανακοινώσεις ως πρόεδρος πρώτον της συστάσεις των συντονιστών στη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου συμφώνησαν οι συντονιστές να μην καταρτήσουμε γνωμοδότηση για την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινή πολιτικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΚΕΠΑ. Στις 4 Σεπτεμβρίου επίσης συμφωνήσαμε να μην γνωμοδοτήσουμε για την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμού για την απαλλαγή του προϋπολογισμού 2016, άλλη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την συνέχεια που ε, δίνεται στην απαλλαγή του οικονομικού έτους 2015 και την έκθεση τη Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και την καταπολέμηση απάτης. Άλλη ετήσια έκθεση είναι αυτή. Στη συνέχεια, ξέρετε ότι συνεδρίασαν ε, σήμερα οι συντονιστέ. Να σας ενημερώσω εν συντομία. Συζητήσαμε την έκθεση για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και ε, ιδρυμάτων. Ορίστηκαν συγκεκριτές η κυρία Μπρέσο με τον κύριο Βίλαντ, σοσιαλιστές δημοκράτες και ΕΛΚ μαζί. Συζητήσαμε συνέχεια την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, στην οποία θα επανέλθουμε όσο νούπο, τη συνεχιζόμενη διαδικασία για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να σταματήσει, είναι δική μου έκθεση αυτή και με επιβεβαίωσαν οι εισηγητή στην νομοθετική πρόταση που θα φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή θα προτείνει ένα κείμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα κάνουμε άλλη νομοθετική έκθεση ίδιας πρωτοβουλία. Και η Επιτροπή μας θα εκφράσει την έντονη αντίρρησή της για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοίμασε και ανακοίνωσε τη νέα της πρόταση αποστολές και ad hoc επισκέψεις στο πρώτο εξάμεινο του 2018 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες ΕΟΧ και υποψήφιες χώρες. Προφανώς θα πρέπει να εγκριθούν αυτές οι αποστολές, αλλά σχεδιάζουμε να πάμε στην Ιρλανδική Δημοκρατία και στο Μαυροβούνιο, ε, το οποίο είναι, όπως γνωρίζετε, υποψήφια χώρα. Ad hoc αντιπροσωπείες τώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ελβετία και Βοσνία-Ζεγοβίνη που δεν είναι ακριβώς υποψήφια χώρα, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει. Ε, ακροάσεις για το πρώτο εξάμεινο του 2018, μια ακρόαση για ε, κοινή επικράτεια, εκλογική, υπερεθνικά ψηφοδέλτια κτλ. Το δεύτερο, ε, δεύτερη ακρόαση ε, σχέση και διαφορά νομιμότητας και νομιμοποίησης, legality και legitimacy. Και το τρίτο, ε, παγκοσμιοποίηση ε, με βάση τις ιδέες του Ρόντρεκ. Ποιος είναι αυτός ο Ρόντρεκ? Α, κατάλαβαν. Και τα μια πρόταση για το ρόλο των πόλεων στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταλλαγή απόψε ενδεχομένω στις 11 Οκτωβρίου με τους Προέδρους ε, της Επιτροπής Περιφερειών Eurocities και τους δημάρχους, το Δήμαρχο της Γάνδης και έναν καθηγητή του ε, Πανεπιστημίου του Ζεσούφ από τη Νοτιοανατολική ε, Πολωνία. Αν δεν διαφωνείτε, προχωρούμε λοιπόν στη μερισσία διαταξή μας, την οποία να βρω όλες. Το σημείο 12 στην ημερήσια διάταξη αφορά την εφαρμογή του Χάρτη Θερμιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σπινέλη. Ρελατρίτσε νομίζω το λένε αυτό στα Ιταλικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές και του ηγητές για την γνωμοδότηση για την αντάλλαγη απόψεων που έγινε στην πρώτη συνεδρίαση του Σκιαδών που έγινε σε 6 Ιουλίου στο Στρασβούργο. Όπως προβλεπόταν να γίνει εκεί, θέλω να επαναλάβω ότι έχω πρόθεση να δεχτώ τη συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την ε, προετοιμασία της, ε, του κειμένου. Όπως τα γνωρίζετε, οι εφαρμοστικές αυτές εκθέσεις με τη διαφορά των συνηθισμένων εκθέσεων πρωτοβουλίας αποτελούνται από δύο μέρη. Ένα που περιγράφει και αναλύει το θέμα που συζητείται και αναλύεται και το άλλο τμήμα είναι περισσότερο πολιτικό, περιέχει τα πολιτικά συμπεράσματα και τις διάφορες συστάσεις για μια βελτίωση, αν αυτό είναι απαραίτητο, της τρέχουσης καταστάσεως η σύνταξη του κειμένου ακολουθεί διαφορετικές δυναμικές και απαιτεί ε, διάφορες δραστηριότητες ε, συμπληρωματικές σε σχέση με τις εκθέσεις πρωτοβουλία συνηθισμένες. Το πρώτο τμήμα θα απαιτήσει έρευνες υπό τη μορφή αποστολών και συναντήσεων με θεσμικούς ε, εκπροσώπους διαφόρων, να οργανώσουμε διάφορες διασκέψεις και εργαστήρια. Μετά θέλουμε και επιστημονική συνεισφορά που θα παρασχεθεί από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου ο, όπως η νομική υπηρεσία και το υπηρεσία μελετών του Κοινοβουλίου και θα ετοιμαστεί ένα έγγραφο εργασίας που θα συνταχθεί ευθύνη της εισηγητρίας και μετά θα συμπεριληφθεί βάση των διαφόρων δραστηριοτήτων που απαιτούνται. Η πρόταση ψηφίσματος λοιπόν θα συνταχθεί ε, βάσει των ερευνών και ε, των στοιχείων που θα συλλεχθούν. Γι' αυτό μια εφαρμοστική έκθεση συνήθως έχει διάρκεια σε ένα έτος. Θα ήθελα ήδη από τώρα να ζητήσω μια ενδεχόμενη παράταση γιατί έχουμε τις διακοπές, στις διακοπές μάλλον καθυστερήσαμε να αρχίσουμε και έχουμε πάρα πολλούς φακέλους, μεγάλος όγκος υλικού προς εξέταση και άρα θα είναι δυσχερέστατο να βρούμε χρονοθυρίδες κατάλληλες ούτως ώστε να καλυφθούν όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες. Πριν εν γέννη να παρουσιάσω το περιεχόμενο, το πολιτικό της εκθέσεως, θα ήθελα εν συντομία να παρουσιάσω το ιστορικό, το υπόβαθρο, ξεκινώντας από το δικό μου όραμα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα η έγκριση του χάρτη εκπροσώπησε κατά την άποψή μου ένα, μια καμπή στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ένωση επισήμως ανέλαβε ευθύνη έναντι των πολιτών της και μεταμορφώθηκε από μια κοινότητα δικαίου σε ένωση δικαιωμάτων. Το άρθρο 6 της συνθήκης εκ των πραγμάτων έδωσε επίσημη συνταγματική σε αυτή την επιλογή και είναι η πρώτη πράξη, αν θέλετε, έναντι επίτευξη άλλων στόχων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ε, τα θεσμικά όργανα ε, εγγυώνται τη συμμόρφωση με τι υποχρεώσει. Ο χάρτη δεν είναι μια απλή διακήρυξη αρχών, προσανατολισμών και αξιών αφηρημένων, αλλά είναι το κανονιστικό θεμέλιο, ε, το απαραίτητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαραίτητη απαραίτητο μέτρο αναφοράς για όλα τα μέτρα που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή που μέτρων που εφαρμόζονται από την Ένωση. προσωπικός πώς θεωρώ ότι ο χάρτης αντιπροσωπεύει ακόμα σε πολλές περιστάσεις ένα μεγάλο, ε, κάποια μεγάλη απουσία. Οι επιλογές ε, που ελήφθησαν επί χάρτου δεν έχουν αποκτήσει πιο ουσιαστική μορφή. Έχουν, υπάρχουν πολλές πολιτικές πρωτοβουλίες που είναι διακυβερνητικές και όχι κοινοτικές Άρα δεν είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις και οι προσανατολισμοί. Δεν επιβάλλονται το κοινοτικό νόμο. Ένα παράδειγμα είναι η πολιτική λιτότητα οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν, διαθετήθηκαν, εφαρμόστηκαν και όχι πάντα μέσω της κοινοτικής μεθόδου. Άρα δεν συμμερίζονται όλοι απόλυτα αυτή τη δική μου αξιολόγηση, το ξέρω αυτό. Θα δούμε καθοδόν πώς ε, θα συμπλέψουμε τελικά και θα πλησιάσουν οι θέσεις μας. Υπό το φως της, της πραγματικότητας ε, θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν την έκθεση. Λοιπόν, θέλουμε να καταλήξουμε σε καλύτερο ορισμό σε επόμενο έγγραφο που θα αντιπροσωπεύσει την βάση από την οποία θα γίνει η ανάλυση. Πάνω απ' όλα, ποιος είναι ο σκοπός της εκθέσεως, ο στόχος. Βασικός σκοπός είναι η ανάλυση της εφαρμογής και εμβέλεια του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, που θα είναι ένα μέσο πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης και ε, δυνάμει το άρθρο 6 των συνθήκων, 6-2 ε, θα πλαισιώνεται από τις συνθήκες. Άρα θα είναι χαρακτήρα αύκο ε, συνταγματικού χαρακτήρα, θεσμικού χαρακτήρα. Τα θεσμικά όργανα και οι φορείς της Ένωσης ε, θα κάνουν την ανάλυση και θα είναι και αποδέκτες των διαφόρων διατάξεων της, ε, του χάρτη. Άρα αποκλείονται τα κράτη-μέλη μεμονωμένα, αλλά μόνο υπό το σχήμα του ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή Συμβούλιο της Ένωσης. Η αξιολόγηση των διαφόρων κρατών μελών αποτέλεσε ήδη αντικείμενο συγκεκριμένων εκθέσεων του Κοινοβουλίου και δεν θα επαναληφθεί αυτή η εργασία. Παραλλήλα θα αποκλειστεί η εμβάθυνση των ενιαίων ε, νομοθεσιών. Θα αναλυθεί ο χάρτης σαν ένα εργαλείο νομικό, πρωτογενούς δικαίου, ε, σφαιρικά επικεντρωνόμενοι επί της λειτουργίας της ρυθμιστικής ε, και κανονιστικής του χάρτη. Πρόθεσή μου βέβαια είναι η εμβάθυνση αντιθέτως της διατάξης του χάρτη αυτού, της χάρτας, άρθρα 51 και 52, που αφορούν την εμβέλεια, το πλαίσιο και την ερμηνεία ε, που απαιτούνται για την εφαρμογή ε, των επιταγών της χάρτας. Στο άρθρο 51 αναφέρονται τα εφαρμοστικά όρια που συχνά επικαιροποιούνται από την ομολογία του ΔΕΚ. Στο άρθρο 52 μπαίνουμε στην ουσία των δικαιωμάτων και των αρχών που αναφέρονται περισσότερο στα άρθρα 51.1 και επιμένουμε επί της ανάγκης να υπάρξει σχέσεις και με άλλα μέσα προστασίας των δικαιωμάτων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι προδιαγραφές και οι συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών. Αφετηρία της αναλύσεως θα είναι η περιγραφή και αξιολόγηση των υφισταμένων μέσων, μηχανισμών και συστάσεων που θετήθηκαν από τα βασικά θεσμικά όργανα της Ένωσης, ούτως ώστε να εφαρμοστεί η χάρτα και να εξασφαλίζεται ο σεβασμό αυτή. Όσον αφορά τα βασικά θεσμικά όργανα της Ενώσης, τέσσερα θα είναι τα πλαίσια και οι τομείς της έρευνας. Η νομοθετική διαδικασία και λήψος αποφάσεων. Σύμφωνα με την οικονομική, δεύτερον, η οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης, τρίτον, η εξωτερική πολιτική και η, πολιτική, η κοινή πολιτική ασφάλεια, τέταρτον, η σημασία που έχει σε εμπορικές συμφωνίες η χάρτα που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Δεν θα μπούμε επί τη ουσία των συγκεκριμένων πολιτικών που υθετούνται από την Ένωση, αλλά θέλουμε να αξιολογήσουμε κατά περίπτωση την εμβέλεια και τη σημασία που έχει η χάρτα σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τους τέσσερις προαναφερθέντες τομείς. Άλλος ενδιαφέρον τομέα έρευνας, κατά την άποψή μου, θα είναι τη εφαρμογής της χάρτας από πλευράς των διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών της Ενώσεως αξιολογούμε ακόμα όσον αφορά αυτό το πόσο είναι φυκτό να γίνει κάτι τέτοιο. και συσχετισμός με τους οργανισμούς αυτούς, διότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ε, και κατανάλωση χρόνου που δεν ξέρω αν έχουμε στη διάθεσή μας. Τέλος, και άλλα δύο θέματα που θα ήθελα να αναπτύξω στην έκθεση. Πρώτο θέμα, η διάδραση μεταξύ διατάξεων της χάρτας και εφαρμοστικών διατάξεων, γενικών εφαρμοστικών διατάξεων που απορρέουν από τη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα άρθρα από το 8 ως 17, ο ρόλος της χάρτας στην προώθηση των στόχων της Ενώσεως και υπό το φως των ορίων που τίθενται από την εφαρμογή των κανόνων αυτών. δεύτερον, η σχέση μεταξύ χάρτας και ηθαγένειας της Ένωσης βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συμμετοχής. Η πρόθεση και όχι μόνο σεβασμός των δικαιωμάτων αντιπροσωπεύει κατά την άποψή μου ένα κίνητρο για τη δημιουργία ενός δημόσιου ευρωπαϊκού χώρου ή του Δήμου, του Ευρωπαϊκού Δήμου όπως αποκαλείται. Μπορεί η χάρτα να είναι ένα από τα μέσα που μπορεί να οδηγήσει στη συμμετοχή των πολιτών μέσω της εγγύησης της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων και της δυνατότητας δικαστικής νομικής επανόρθωσης προβλημάτων. Για να υπάρχει καλύτερη επάσπαση αυτών. Όπως είπα στην αρχή, θα ήθελα αυτή η συνεδρίαση να είναι το πρώτο βήμα για μια κοινή διαδρομή συμμετοχική και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για όλες τις απόψεις ε, και προτάσεις που μου κάνετε ήδη από σήμερα και μέσω ανταλλαγών μέσω της γραπτής διαδικασίας και μέσω μελλοντικών συναντήσεων. Κάθε δική σας συνεισφορά για μένα θα είναι χρησιμότατη. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στους Ε, Δεν είναι κανείς εδώ βεβαίως. Ε, έχω ένα έγγραφο από τον Έλμαρ Μπρόκ που μου ζήτησε να διαβάσω και θα το διαβάσω. Αγαπητοί συναδελφοί, δυστυχώ δεν μπορώ να έρθω συνεδρίαση απόψε. για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου και μετά μου ζητάει να πω λίγα λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μάργαρα Σπινέλη που παρουσίασε την ε, δομή και το χρονοδιάγραμμα πριν από τη συνάντηση του Στρασβούργου. Και ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι και αρμοδιότητες άλλων επιτροπών του Κοινοβουλίου, όπως σωστά ανέφερε η η Μπάρμπαρα. Πρέπει να συμφωνήσουμε στην προσέγγιση στο πεδίο εφαρμογή και στην ουσία. Όπω πάντα βεβαίω ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Οπότε πρέπει να έχουμε μια λεπτομερή πρόταση σύντομα και θέλω να τονίσω την ανάγκη να συζητηθεί το πεδίο εφαρμογή του άρθρου 51 και παραπέρα εκεί όπου το Brexit μπορεί να δώσει περαιτέρω όθηση. Αναμένω τις προτάσεις σας και σας ευχαριστώ για την προσέγγιση αυτή που επιλέξατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Κάποια άλλη ομάδα θέλει να προσθέσει κάτι, όχι. Ναι, ναι, καλώς μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Σίρβια Κόφμαν, η σκιώδης μας, απουσιάζει. Και αντίθετο συνάδελφο Μπροκ δεν μου έδωσε ακόμα κάποιο κείμενο να διαβάσω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα Σπινέλη για αυτή την παρουσίαση, την διεξοδικότατη. Θα ήθελα να πω ότι η τοποθέτησή της θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. θα μας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε και να συμβάλλουμε στον αφορά την τοποθέτησή της. Και μετά η συγκήτριά μας Σκιώδης θα, θα εξηγήσει καλύτερα τη συνεισφορά μας. Πιστεύω ότι κάποια θέματα που παρετέθησαν στο έγγραφο που μόλις τώρα μας επενθύμισε η Μπάρμπαρα Σπινέλη είναι ενδιαφέροντα θέματα. Βλέπω ότι υπάρχει δυνατότητα εφαρμογή αυτών των αρχών. Δημιουργούνται πιθανότητες. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι ζητείται εμβάθυνση πρέπει να αναλύσουμε αν μπορεί να εφαρμοστεί να εφαρμόσει και συλλογικά δικαιώματα η χάρτα και όχι μόνο ατομικά. Άρα να διευρύνουμε κάπως την κάλυψη. Να υπάρχουν και γενικότερες εγγυήσει, όχι μόνο ατομικές για τους πολίτες. Πιο συλλογικές, πιο ομαδικές. Διερωτώ με. Μήπως ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα πεδία. Ενδιαφέρον το θέμα των οργανισμών και των υπηρεσιών της Ενώσεως αυτή τη στιγμή δεν θα είχα απάντηση προς εξερεύνηση του θέματος. Θα ήταν ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε και κάποιες φορείς και οργανισμούς διότι θα εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς. Πώς ενδεχομένως θα μπορέσουμε να διαβρύνουμε το πεδίο που θα καλύπτεται από τη χάρτα. Εκτός αν μου διέφυγε, έχω κάτι άλλο να θέσω. Άλλα ζητήματα. Όπως τα προβλήματα που δημιουργεί το Brexit. Πώς εφαρμόζονται, Φερρυπίν, τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα προστατεύονται, πώς θα τα εγγυηθούμε. Σε μετανάστες επίσης, πρόσφυγες. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ή εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως θεωρείται η εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων αυτόματη και αποτελεσματική και ουσιαστική. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλο ενδεχόμενο πεδίο εφαρμογή που θα ήταν ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ αυτά που αναφέρατε ήταν ενδιαφέροντα ζητήματα διότι διευρύνουν κάπως την προοπτική, τις προοπτικές εφαρμογής της χάρτας και θα μπορούσαν να βοηθήσουν επεξεργασία μελλοντικών, εν ώψη μελλοντικών συνθήκων να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένας από τους στόχους που θέτει η εισηγήτρια, αλλά και ένας στόχος που θα πρέπει να θέσουμε συνολικά σαν Επιτροπή. Ευχαριστώ εν τω μεταξύ. Οι σκιώδεις μας θα είναι ευτυχής να συνεργαστεί μαζί σας, είναι σίγουρο. Thank you indeed. Ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Καλά, δεν είστε και υποχρεωμένοι, άμα δεν θέλετε. Όχι, όχι, είμαι στην διάθεσή σας, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Εκτός από αυτό δεν έχω κάποια συγκεκριμένη συνεισφορά. Απλά να πω ότι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την δουλειά που γίνεται. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Επ' αυτού νομίζω. Οπότε πάμε στο τελευταίο ουσιαστικό θέμα που αφορά εμένα. Είναι ο κανονισμός ε, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Λοιπόν, Είχα γράψει εγώ την έκθεση που ψηφίστηκε πριν από δύο χρόνια. Δεν είναι νομοθετική έκθεση. Ε, ήταν έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας με στόχο να βελτιωθεί ο κανονισμός 21-20-0211. Ε, Δεν συνέβη τίποτα ιδιαίτερο. Μάλιστα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στα πρακτικά των επιτρόπων το περιέγραψαν ως κάτι το επικίνδυνο Εν τω μεταξύ, κάπου 60 τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει. Ούτε μία δεν έχει επιτύχει. Οπότε ο στόχος από τη δική μας τη Σκοπιά ήταν να προσπαθήσουμε το μέσο αυτό να λειτουργήσει. Να μεταφέρει τις επιθυμίες των πολιτών προς την Κομισιόν με στόχο να βελτιωθεί η νομοθεσία. Μετά, φέτος το καλοκαίρι, ξεκινήσαμε την νομοθετική πρωτοβουλία, μια έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας, πάλι εγώ εισηγητής, με στόχο φέρουμε σοβαρές αλλαγές στην 21-20. Μετά, δεν ακούσαμε τίποτα από την Κομισιόν, μετά με κάλεσε ο κύριος Τίμερμανς μαζί με τους εισηγητές, τους κυρίους Τζαμπάσκι και Βαλέσα, και τότε με ενημέρωσαν ότι δεν θα ήταν αλλαγή, αλλά μεταρρύθμιση εν ολίγης ένας νέος κανονισμός. Κάποιοι εξεπλάγησαν και λίγες μέρες μετά εμφανίστηκε ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά είναι ένας νέος κανονισμός. Και από ό,τι αντιλαμβάνουμε η Κομισιόν θέλει να ε, πέρασει από όλα τα στάδια της διαδικασίας και να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020. Οφείλω να πω ότι το έγγραφο αυτό με τις μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μας εξέπληξε. Δεν μας έδωσαν κάποιες πληροφορίες. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η δουλειά που έχουμε κάνει πλέον είναι πέριτη και νομίζω εδώ πως πρέπει να πω ότι η διοργανική συμφωνία προβλέπει τα εξής. Η Συμφωνία Πλαίσιο προβλέπει ότι η Κομισιόν θα λάβει υπόψη τις απόψεις Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, ειδικά σε σχέση με την βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης. Δεύτερον, η Κομισιόν δεσμεύεται να εμπλακεί σε επικοδομητικό διάλογο, να βελτιώσει την ροή πληροφοριών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, να βελτιώσει συνεργασία μεταξύ των οργάνων και να βελτιώσει τον σχεδιασμό και την, τον συντονισμό. Τρίτον, ε, μπορεί να γίνει, γίνεται μια αναφορά στην παράγραφο 13 που λέει πως η Κομισιόν δεν θα δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση ή σημαντική απόφαση ή πρωτοβουλία πριν ειδοποιήσει γραπτό στο Κοινοβούλιο. Και βεβαίως ε, να υπενθυμίσω και την επιστολή της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών που επισήμως ε, ανακοίνωνε την σύνταξη της έκθεσης αυτής ε, προς την Κομισιόν. Οπότε, έτσι έχουν σήμερα τα πράγματα. Σήμερα οι συντονιστές αποφάσισαν ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τη δουλειά που είχε γίνει στην προηγούμενη έκθεση, την 2.11, ε, και θα ξεκινήσουμε μία νέα έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας ε, επί τη φάση του εγγράφου που έχει δημοσιεύσει η Κομισιόν. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν υπερβάλλω νομίζω όταν λέω ότι υπάρχει σοβαρή δυσαρέσκεια εντός της Επιτροπής μας, δεν το λέω μόνο εγώ. Πολλοί θεωρούμε ότι η Κομισιόν δεν μας μεταχειρίστηκε δίκαια. Αυτή είναι η θέση μου. Έναν άλλο συνάδελφο βλέπω μόνο εδώ, την Μπάρμπαρα. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε και εσείς κάτι, αλλιώς θα δώσω λόγο στην Κομισιόν αν έχουν και αυτοί να πούν κάτι. Θέλετε να κάνω παρέμβαση κανονική. Ό,τι θέλετε να πείτε. Καταρχάς, στα αγγλικά η κυρία Σφινέλη, θα ήθελα να πω το εξής. Συμφωνώ πάρα πολύ με την δυσαρέσκειά σας ε, ως προς τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ρόλος όσο και η σημασία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων δεν ε, αξιολογήθηκε σωστά, ούτε όλη ε, η δουλειά που έχει κάνει και ο κόπος του εισηγητού για το θέμα αυτό. Επιτρέψτε μου να τονίσω μερικά σημεία ε, για την πρωτοσία. Θα πω στα Ιταλικά όμως. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ζητήματα κρισίμου σημασίας κατά την άποψή μου τα οποία δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που συζητήθηκαν ήδη από το 2015 στο, στην έκθεση Σέφλιν και αναφερόνται στην έκθεση και συζητούντο. Στη δεύτερη έκθεση που αναφέρθηκε, η οποία ολοκληρώθηκε. Ένα σημείο θεμελιώδης από αυτά του κανονισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη δύο αποφάσεις του ΔΕΚ στην επιχειρηματολογία όσον αφορά τι πρωτοβουλίε των πολιτών. Safe Pack και TTIP, δηλαδή τη δυνατότητα να παρουσιάζονται πρωτοβουλίε ε, για ειδήποτε νομοθεσία, νομοθετική πράξη. Δηλαδή, η ανάγκη σαφέστερου ορισμού τι σημαίνει το legal act, μια νομοθετική πράξη. Για το δικαστήριο είναι πιο εκτεταμένη η ερμηνεία από αυτή που ε, παρουσιάζεται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλο σημείο που δεν καλύπτεται είναι το αίτημα του Κοινοβουλίου που έγινε το 2015 να προβλέπεται υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει νομοθετική πράξη εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος σε απάντηση μιας πρωτοβουλίας ε, πολιτών που έγινε αποδεκτή. Επ' αυτού και επί άλλων σημείων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα υπερασπίστηκε με ζήλο την εξουσία ε, την πρωτοβουλία που έχει, το δικαίωμα πρωτοβουλίας, που πρέπει με καχυποψία να δει κανείς την εμβέλεια αυτής της τάσης. Είναι το εργαλείο που βλέπετε από το άρθρο 11 των συνθήκων, που είναι δεσμευτικό όμως για τα θεσμικά όργανα. Κάτι άλλο. Ο κανονισμός δεν αναφέρεται στο θέμα του διπλού ελέγχου από πλευράς... Ευρωπαϊκής Επιτροπή και τη στιγμή της καταχώρησης της πρωτοβουλία, κατάθεση πρωτοβουλίας... και εξετάζοντας την πρωτοβουλία όταν έχει ε, συλλέξει ένα εκατομμύριο υπογραφές. Και αυτό είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την τάση να μονοπολεί όλη τη διαδικασία. Και αυτό αφορά κυρίως το θέμα των δημοσίων ακροάσεων. Αν θυμάμαι σωστά, όπως αναφέρθηκε από τον η ακρόση θα έπρεπε να είναι που θα διοργανώνεται με ουδέτερο τρόπο από το Κοινοβούλιο αλλά όχι από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για άλλη μια φορά υπάρχει προσπάθεια μονοπολίσεως του θέματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατά την άποψή μου δεν είναι καθόλου σωστό σαν προσέγγιση. δεν είναι ορθό και η Επιτροπή ΑΦΚΟ, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να καταστήσει αυτές τις ακροάσεις πιο ανεξάρτητες. Το 2015 η διοργάνωση δημοσίων ακροάσεων έπρεπε να εξάγεται υπό την αιγίδα ουδέτερης επιτροπής που να, είναι, να μην είναι η διαρμόδια για το θέμα αυτό που αφορά η πρωτοβουλία των πολιτών. Σταματώ εδώ και ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλει κανείς να λάβει το λόγο, να προσθέσει τίποτα. Or is it still silence? Επικρατεί σιωπή. Ε, καλησπέρα σας. Ε, περιμένουμε, να περιμένουμε πέντε λεπτά το τμήματάρχη να έρθει ε, στην ε, συνεδρία. Δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί, είναι καθοδόν. Well, as you asked nicely, the answer... Να περιμένουμε πέντε λεπτά αφού το ζητάτε τόσο ευγενικά, αλλά μόνο πέντε λεπτά, γιατί είναι πολύ προχωρημένη η ώρα και πέμπτη απόγευμα, πεντά λεπτή διακοπή και θα επαναλάβουμε παρά είκοσι. Ναι, ευχαριστώ πολύ λιγότερο από πέντε λεπτά. Ορίστε, κατέφτασε. Μάλιστα. Άρα επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση. I'm sorry. Διαδικαστικό η κυρία Σπινέλη. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω, μάλλον να το πω αλλιώς, λυπάμαι πάρα πολύ για την καθυστερημένη άφηξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνεδρίαση αυτή. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν άκουσε καν τις αντιρρήσεις μας. Προτείνεται ένας κανονισμός εδώ, με τρόπο ευνηδιαστικό, διακόπτοντας ε, τις εργασίες του εισηγητού μας για το θέμα αυτό και ακόμα και σε τούτη εδώ τη συνεδρίαση ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται κατόπιν εορτής αφού παρουσιάσαμε εμείς το θέμα πραγματικά έχω μπουχτίσει με τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα κανονικά παρατέταρτο ξεκινούσε αυτό το θέμα, οπότε έχει δικαιολογία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αρχίσαμε την εξέταση του θέματος αυτού νωρίτερα. Αλλά επειδή διεκπαιρεώσαμε τόσο γρήγορα τα θέματα, γι' αυτό. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Good afternoon and indeed. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα πριν ζητήσω συγγνώμη να συστηθώ αλλά περιμέναμε να συζητηθεί το θέμα αυτό παρατέταρτο. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν και είπα να πλύνω και τα χέρια μου, γι' αυτό άργησα. Ρούτι και Μπόγκερτ λέγομαι, τμήματάρχης, υπεύθυνο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Βεβαίω καλύπτουμε και άλλα θέματα, τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους Χαίρομαι λοιπόν που ήρθα εδώ, ίσως ε, όχι υπό τις καλύτερες ε, συνθήκες, αλλά ανέλαβα τον Ιούλιο, πολλά πράγματα έχουν συμβεί έκτοτε και τα γνωρίζουμε όλοι και βεβαίως ε, θα συμβούν και στο προσεχές μέλλον για να επιτύχουμε τον στόχο μας, δηλαδή να βρεθεί μια κοινή συμφωνία με τους συνομοθέτες. Λοιπόν, έξω την εισαγωγή, δεν ξέρω σε τι ακριβώς θέλετε να εκφέρω απόψε. Πείτε μου. Σας καλωσορίζω κύριε Μπόχαρτ στην Επιτροπή. Νομίζω εκφράσαμε την δυσαρέσκειά μας. Αρχίσατε να ζητάτε κάποια συγγνώμη. Εάν έχετε να προσθέσετε κάτι σε σχέση με το πώς βλέπετε τα πράγματα στο μέλλον. Και αν έχετε κάτι να πείτε για την απόφαση δηλαδή να σταματήσουμε με την προηγούμενη έκθεση και να ξεκινήσουμε μια καινούργια. Και νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο θεσμικών οργάνων να υπάρχει μια σωστή πληροφορία, ροή πληροφοριών από εδώ και μπρος. Θα είμαι ήπιος, αλλά κάποιοι συναδελφοί μου είναι εξοργισμένη για το ότι σταμάτησε η ροή των πληροφοριών. Αυτό παραβιάζει και την διοργανική συμφωνία. Οπωσδήποτε στο πνεύμα και ίσως και το γράμμα της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Ίσως καλύτερα που μου διέφυγε η η διέκφρασή της δυσαρέσκειάς σας. Ε, μπορείτε να το δείτε πάντα στο διαδικτύο. Λοιπόν, Πρώτα απ' όλα γεγονός, ε, αναγνωρίζω πράγματι ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια και είναι και κατανοητή. Εγώ βεβαίω είμαι υπάλληλος Κομισιόν, εκπροσωπώ την θέση του Σώματος των Επιτρόπων και εκεί θα μείνω. Υπήρχε ήδη μια συνάντηση σχετική και ήδη ο πρόεδρο τη Επιτροπή Δεγματικών Δημάτων έχει εκφράσει την άποψη αυτή και υπήρξε μια πρώτη απάντηση. Αντιλαμβάνομαι ότι και επίση ο Επίτροπο θέλει να λειτουργήσει το θέμα αυτό και η πρόταση αλλά και βεβαίως η συνεργασία με το Κοινοβούλιο και θέλει να συνεχίσουμε και τις συναντήσεις όπως είχαμε στο παρελθόν οπότε αντιλαμβάνουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση τώρα δεν θα σας πω εγώ αν είναι η κατάλληλη στιγμή να εκφραστείτε αλλά είστε σίγουρα σοφός άνθρωπος ε, αναγνωρίζουμε ε, εμείς που καθόμαστε εδώ την κατάσταση ως έχει και αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ και ήδη ήρθα σε επαφή και με τη γραμματεία είναι να έχουμε μια όσο δυνατόν πιο γρήγορη και ταχεία ροή πληροφοριών. Ε, να σας πω, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη στιγμή να το πούμε, η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να οργανώσει όπου και όποτε θέλετε μια ακρόαση γιατί υπάρχουν κάποια σχετικά στοιχεία. Δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να διατρέξετε το έγγραφο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς όπου καλό είναι να ενημερώσουμε πριν ξεκινήσει η συζήτηση και είμαστε έτοιμοι μόλις μας πείτε ε, με τους ανθρώπους που θέλετε εσείς ε, γιατί φαντάζομαι θα είναι παραπάνω από μια επιτροπή που θα εμπλακεί. Θα έρθουμε σε επαφή με τις γραμματείες ε, ακριβώς για να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα. Ελπίζω όσοι έριξαν μια ματιά στην πρόταση να είδαν ε, ότι δεν αγνοήσαμε το ψήφισμα του 2015 ούτε την ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας Ελπίζω ότι θα βρήκατε αρκετά στοιχεία τους εκεί μέσα και θα είστε ικανοποιημένοι. Πάντα βεβαίως κάποια στοιχεία παραλείπονται και ελπίζω μετά να έχουμε νομίζω μια σωστή διαβούλευση. Ε, μπορούμε να επανέλθουμε εδώ ή υπό κάποια άλλη σύνθεση για να εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, πολύ. Καλά, δεν είπα ακριβώ αυτό, κάτι κοντινό. Βεβαίως ε, δεχόμαστε την προσφορά σας για ε, περαιτέρω ε, μια σύσκεψη εργασίας, ας πούμε, νομίζω είναι μια καλή ιδέα. Έχουν μείνει μερικά μικρά θέματα. Να προσθέσω ότι αν θέλετε πραγματικά να ακούσετε τη δυσαρέσκειά μας, θα τα πω στα ογκρικά. Αλλά ευτυχώ ε, τη γλιτώσατε, διότι δεν έχουμε διερμηνία από τα ογκρικά, αλλιώς θα τα ακούγατε. Και αυτό <laughs> θα σα ε, ε, έπιθε μάλλον. Λοιπόν, στα διάφορα, Μπάρμπαρα, έχεις κανένα διάφορο, γιατί δυο μα έχουμε μείνει. Όχι, νομίζω αυτό ήταν η απάντηση. Επόμενη συνεδρίαση. 11 Οκτωβρίου, συμφωνούν τα έγγραφα μάλιστα, στις 9 το πρωί και στη συνέχεια στις 2.30 το απόγευμα, το μεσημέρι, στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της. Λήξη συνεδρίασης και μπορούμε όλα να πάμε στα σπίτια μας με το καλό.